liebe Kolleginnen und Kollegen. Θα πρότεινα λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να συνεχίσουμε τη απογευματινή μας συνεδρίαση. Πριν περάσουμε όμως στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να σας πω ότι ο συνάδελφος Κρίστεσεν έχει ένα τηλεοπτικό συνεργείο ε, που ε, το ε, Μαγνητοσκοπή, τραβάει πλάνα. Ε, σα το λέω για να το ξέρετε. Το δεχόμαστε, είναι εγνώση μας. Ε, περνάμε λοιπόν στο σημείο 9 της σα διάταξης. Εκφράστηκε η επιθυμία από την Επιτροπή μας να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διάφορες γενικές διευθύνσεις ε, γεωργία ανταγωνισμού και εμπορίου σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ευρωπαϊκού τομέα βοήου κρέατος. Η συζήτηση λοιπόν αφορά το Μερκοσούρ και την εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και πέρα από αυτό. Να δούμε γενικά το τομέα του βαϊού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρεις εκπροσώπους έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Πολ Σουσάχ, ελπίζω να μην κατακρεωργώ το όνομά σας. Ε, Διευθυντή στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, ανταγωνισμού, συγγνώμη, κύριος Μάικλ Σκάνερ, στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας εκτελεί χρέη αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού και την κυρία Κοντούνη, ε, που είναι τμήματάρχη στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. θα σας παρακαλούσα ε, να λάβετε το λόγο για 20 λεπτά συνολικά. Συνεννοηθείτε μεταξύ σας παρακαλώ με ποια σειρά. Εδώ στο δικό μου πρόγραμμα βλέπω ότι θα λάβει πρώτος ε, το λόγο ο κύριος Ισάρα από τη Γενική Διεύθυνση Συνταγωνισμού. Ε, Ή ο κύριος Κάνελ. Δεν ξέρω, κανονίστε το μεταξύ σας. Συνολικά περίπου 20 λεπτά παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά να μπορώ να σας ενημερώσω για την κατάσταση της αγοράς του βοήου και των προϊόντων βοηδού. βοηδούς. Να ενημερώσω ότι αυτή την κατηγορία προϊόντων δεν μπορούμε να τη δούμε και απομονωμένη βεβαίω, αλλά στο πλαίσιο του τι συμβαίνει στην αγορά με τα ζωικά προϊόντα γενικώ. Η αγορά, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πολύ ε, ευάλωτη ε, και ε, ευπαθής ως προς τις διακυμάνσεις. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε τη σταθερότητα και τους κοινοτρόφους μας από διάφορους τρεγμούς και κλειδονισμούς που μπορούν να προκύψουν από την αστάθεια στην αγορά. Εάν δούμε τι γίνεται με την αγορά προϊόντων κρέατος, η κατάσταση είναι δύσκολη. Στην αγορά του κρέατος βέβαια τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Σε μεγάλο μέρος του χείριου κρέατο. στην αγορά του χείριου κρέατος πάνε καλά τα πράγματα, ε, λόγω του πανόλη των χείρων στην Κίνα, πράγμα που έχει ανεβάσει τη ζήτηση στα δικά μας προϊόντα. Το μέσο των γαλακτοκομικών στην Ευρώπη επίσης τα πάει σχετικά καλά, αν και δεν είναι στα υψηλά επίπεδα των τελευταίων ετών. Στα πουλερικά επίση τα πράγματα πάνε καλά σε μεγάλο βαθμό λόγω της τάσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ε, παγκόσμιας τάσης να αυξάνεται τη ζήτηση στο κρέας των πουλερικών. Και επειδή η ζήτηση στην Κίνα επίσης έχει περάσει από την ε, ζήτηση για χείριο τα πουλερικά. Στο αρνήσιο, στο εγωπρόβιο κρέας, τα πράγματα είναι σταθερά, ενώ φτάνουμε τώρα στο Βόιο που η κατάσταση αλλάζει σημαντικά. Κατά γενική ομολογία, η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Βόιο Κρέας μπορεί να είναι πηγή ανησυχίας, σοβαρής ανησυχίας. Η πτώση της ζήτησης για το βόιο και τα προϊόντα βοηδούς, οι αλλαγές στους τρόπους κατανάλωσης και στις εμπορικές τάσεις έχουν ακριβώς προκαλέσει αυτό. Επίσης η δομή του τομέα με μικρές εκμεταλλεύσεις, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οδηγεί στην επίταση της κρίσης. Εάν δούμε το βαρόμετρο για την υγεία του τομέα αυτού θα πρέπει να δούμε τις τιμές. Η αντιπροσωπευτική τιμή για τα προϊόντα βόηου βλέπουμε πτώση 4% τους 12 τελευταίους μήνες. Ωστόσο, αυτό υποκρύπτει σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Λόγω χάρη, το κάτω μέλος που είχε τη μεγαλύτερη πτώση στις τιμές είναι η Πολωνία. Οι τιμές έπεσαν κατά ένα 9%. Ακολουθεί η Σουηδία με πτώσεις ε, της τάξης του 7%, η Γερμανία 6,6%, και μετά έχουμε μια ομάδα χωρών, Ιρλανδία, Ενωμένο Βασίλειο και Δανία, με πτώση 5,5 έως 6%. Εάν δούμε τις γενικότερες τάσεις, ένας μικρός αριθμός κρατών μελών, ιδίω η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Γαλλία, κατέγραψαν μικρές περιορισμένες αυξήσεις στις τιμές. Τονίζω ότι οι αλλαγές αυτές τις τιμές έχουν να κάνουν με τα βασικά προϊόντα βόλου ό,τι κατηγορία και να πάρουμε, είναι παρόμοιες οι τάσεις, γι' αυτό παίρνουμε την ε, πιο αντιπροσωπευτική. Βεβαίως για τη δυσχερή κατάσταση στην αγορά υπάρχουν και κάποιες εξηγήσει. Ο πρώτος τομέας που πρέπει να δούμε εδώ είναι οι εξαγωγές. Εκεί βρίσκουμε μέρος της εξήγησης. Οι εξαγωγές είναι περιορισμένες έχουν μειωθεί κατά 4,4% του πρώτου 8 μήνε τη φετινή χρονιά σε σχέση με περασμένα έτη. Και αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντε. Πρώτον, σχετικά οξυμένη ε, μείωση στις εξαγωγές προς την Τουρκία, ζών των ζώων προς την Τουρκία, και κατά συνέπεια επηρεάζεται και το βόλιο. Επίσης, ε, ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι τωρινές δυσκολίες στην αγορά δεν έχουν να κάνουν μόνο με αύξηση στις, εξαγωγές, εισαγωγές. Οι εισαγωγές είναι και αυτές ε, σχετικά μειωμένες, έχουν ε, πέσει κατά 4,7% και σε ένα συνολικό διεθνές τοπίο παραμένουμε ένας μικρός παράγοντας στην αγορά για τα προϊόντα και τα βοηδούς κρέατος. Ε, εάν δούμε τι γίνεται με την αναλογία με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα, έχουμε μια πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σύγκριση με αυτούς. Επίσης, έχουμε ένα εμπορικό πλεόνασμα στους περισσότερους τομείς κρέατος. Το βόλιο πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο της συνολικής αγοράς για προϊόντα ζωικής προέλευσης. Έχουμε πέντε δις λόγου χάρη μα στο χείριο. Σοβαρά πλοενάσματα και για, για τα ζώντα ζώα και για τις ε, ζωοτροφές για κατοικίδια και για τα ε, ε, εντόστια. Αυτά όλα εμέσως στηρίζουν τον τομέα του βοηού. Θέλω λοιπόν να τονίσω και πάλι ότι ο, τομέα μας, ο τομέας μας του βοηού ωφελείται από τη γενική εμπορική ε, τάση και εξέλιξη. Τώρα, ένα άλλο στοιχείο που επηρεάζει το εμπόριο είναι η κατανάλωση. Δεν έχει αλλάξει και βρίσκεται και σε φάση μεταβολής. Τα τελευταία 10 χρόνια η κατακεφαλή κατανάλωση βόηου ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 4,5%. Αυτό από μόνο του δεν φαίνεται φοβερά σημαντικό, αλλά εάν το συγκρίνουμε με τους ανάλογους αριθμούς για το κρέας πουλερικών, η κατακεφαλή κατανάλωση κατακεφαλή κατανάλωση αυξήθηκε κατά 22% για ολόκληρη αυτή την περίοδο. Αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν τριπλάσιο κρέας πουλερικών κατά κεφαλή αντί βόλιο. Αυτά λόγω των συνηθιών διατροφής, ε, των όσων κυκλοφορούν για την υγεία και τις κλιματικές αλλαγές. Έχει μειωθεί και θα μειωθεί περαιτέρω η κατανάλωση βόλου. Αυτό λένε οι προβλέψεις. Βεβαίως παραμένουν προβλέψεις. Αλλά ο ε, ορίζοντας για το βόλιο είναι μάλλον ορίζοντας απεσιοδοξίας. Ε, σε αντιδιαστολή η κατανάλωση παγκοσμίω ε, για το βόλιο προβλέπεται να αυξηθεί έστω και περιορισμένα πάντα σε σύγκριση με το κρέας πουλερικών λόγου χάρη. Ταυτόχρονα η κατανάλωση των νέων εναλλακτικών για το βόλιο έχει κατάσταση αυξητική, αλλά δεν έχει βρει και άμεση δίωδο στην αγορά. Ένας σαφής παράγοντας για τις ε, δυσχέρειες της αγοράς είναι βεβαίως και η κατάσταση αναταραχής λόγω του Brexit. Δεν θα περάσω σε λεπτομέρειες, γιατί όλοι γνωρίζετε τις προβλεπόμενες συνέπειες, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια μεγάλη αγορά εξαγωγών βόηου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε τη σημασία τους και οποιαδήποτε εξαγωγή από τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς εκείνους αποσταθεροποιεί την αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το Brexit και η σχετική πτώση της ε, αγγλική Τερλίνας που έχει πέσει κι άλλο ένα επιπλέον 13-14% σε σχέση με τον καιρό του δημοψηφίσματος το 2016. Έχει πολύ αρνητικές συνέπειες και για την αγορά του βόλου και για τις ε, εξαγωγές και εσωτερικώς. Επίσης, η πιθανότητα ενός Brexit χωρίς συμφωνία που θα έχει να κάνει και με τους δασμούς εξαγωγών μάλλον από τους 27 ε, της Ευρώπης προς το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό αποσταθεροποιεί και οδηγεί σε πτωτική τάση την αγορά. Αυτό ισχύει όλος ιδιαίτερος για την Ιρλανδία που παραδοσιακά είχε πολύ στενούς δεσμούς με την αγορά βόηου του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι λοιπόν οι δυσκολίες της αγοράς βοήου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν να κάνουν και με την παραγωγή, η οποία είναι επικεντρωμένη σε μικρής κλίμακας κτηνοτροφικές μονάδες. 43% 87% στις κάτω χώρες ε, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό με 4% στην ε, Ρουμανία. Αυτό δείχνει ότι οι μονάδες οι μονάδες μεγάλων βοηδών έχουν τάση να συγκεντρώνονται. Ο ανταγωνισ... Τα θέματα ανταγωνισμού επίσης είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την αγορά και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της τον Οκτώβριο του 2018 διερευνώντας το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες ανταγωνισμού στον τομέα ε, τον αγροδιατροφικό το σημείωμα που απευθυνόταν στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και, και συνόδευε την έκθεση είναι εύγλωτο. Από το συνολικό αριθμό μελετών που έγιναν για τον τομέα των βοηδών, ε, οι περισσότερες περιπτώσεις, το 1 τρίτο μάλλον, οδήγησαν σε επιβολή προστήμων. Το τι γίνεται τώρα με τα κράτη-μέλη σε αυτές τις περιπτώσει ε, είναι βασικά ότι έχουμε τέσσερι επιλογέ στρατηγική. Πρώτον, απευθείας πληρωμές από τον πρώτο πυλώνα που επιτρέπουν ένα βασικό επίπεδο υποστήριξης για τις μονάδες που πλήττονται. Αυτό βεβαίως μπορεί να συμπληρωθεί και από τις επιστροφές της αγοράς, των οποίων την αξία δεν μπορούμε να υποτιμούμε, ακόμα και στις σημερινές δυσχερείς συνθήκες για την αγορά. Δεύτερος παράγοντας, η οικειοθελής συνδεδεμένη βοήθεια. Όπως λέμε, είναι θελούσια αλλά στην πράξη χρησιμοποιείται από σημαντικό αριθμό κρατών μελών για να υποστηρίξουν τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους. Ε, και ο τομέας του βόηου είναι το 40% του, της συνολικής ε, πρόσληψης, αποδοχής αυτής της οθελούς συνδεδεμένης βοήθειας, 23 τα που προσφέρουν 7 δις συνολικά βοήθεια στους παραγωγούς βοηδούς. Ένα άλλο στοιχείο είναι τα κονδύλια τη ανάπτυξη τη υπαίθρου των Πολιών 2 με πολιτικά προγράμματα, δράσει υποστήριξη, προσπάθειε έρευνα στην αγορά, νέε επενδυτικέ προσπάθειε και διευκολύνσει και ομάδε παραγωγών που μπορεί να υποστηριχθούν ω προ την αηφορία και τα μέτρα υποστήριξη τη κοινοτροφία. Και μετά τα άμεσα μέτρα υποστήριξη τη αγορά, ένα μέτρο που αφορούσε την Ιρλανδία με 50 εκατομμύρια για 35.000 κτηνοτρόφους στην Ιρλανδία. Το μέτρο αυτό προσήλ... συνάντησε κάποιες αντιρρήσεις από τα κράτη-μέλη, αλλά η Ιρλανδία ήταν το κάτω μέρος που είχαμε υπόψη με αυτό το μέτρο και, τα κάτι και άλλα κράτη-μέλη υποφελήθηκαν. Όπως με τη διευθέτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποτίθεται ότι θα κατέρε αν έρχονταν εκατοντάδε χιλιάδε τόνοι Ιρλανδικού βόηου, αλλά τελικά πήγε προ το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν κατέκλυσε όπω υπολογιζόταν τι ενωσιακέ αγορέ. Ο τομέα γενικώ λοιπόν επωφελήθηκε από αυτό το συγκεκριμένο μέτρο. Και τέλο, πρέπει να τονίσω ότι το βόλιο παρομένει ένα δύσκολο, ένα ευαίσθητο προϊόν στις εμπορικές μας διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μικρός παράγοντας διεθνώς ως προς το βόλιο και τα πρώτα βοηθούς και επιμένουμε στις εμπορικές μας διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας ότι το προϊόν αυτό για μας είναι ευαίσθητο, έχει μια ιδιαίτερη σημασία και έχει σημασία επίσης να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των κοινοτρόφων μας. Ως προς τις μελλοντικέ εξελίξεις και το τι φαίνεται να διαγράφεται στον ορίζοντα. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την Κίνα και την Πανόλη των ε, Χείρων. Εκεί υπάρχει τεράστια έλλειψη στη χώρα αυτή, ε, μειωμένη παραγωγή ε, και συνολικά μικρότερη από τη ΣΥΠΑ και τη Βραζιλία και την παραγωγή τους εγωπρόβιου κρέατος. Αυτό με τις εισαγωγές βοηού δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο. Κοιτάζουν λοιπόν για εναλλακτικές Εκεί ε, μπορεί να παίξει ρόλο το βόλιο και ίσω οι δικοί μα οι εμπορευόμενοι θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Έχουμε δει να επιτελείται κάποια πρόοδο στι τελευταίε εβδομάδε και μήνε ω προ την πρόσβαση στην αγορά τη Κίνα για βασικά για κάποια από τα σημαντικά μας κράτη-μέλη. Αυτό ισχύει και αλλού στην Ασία. Δεν έχει άμεσα σχέση με την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, αλλά υπάρχει θέμα πρόσβαση στην αγορά και στην Νότια Κορέα λόγω χάρη. Κάποια κράτη-μέλη, Ιρλανδία ιδίω, κατάφεραν να πάρουν έγκριση για κάποιε από τι ε, εξαγωγέ του βόλου και νοπού βόλου. Βεβαίω δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δική μα την εσωτερική αγορά. Είπα προηγουμένω ότι παρά τις δυσχερεί μελλοντικέ ε, προβλέψεις υπάρχει και μεγάλη ανισομέρεια μεταξύ της κατακεφαλής κατανάλωσης των κρατών μελών. Λόγω χάρη στη Βόρεια Ευρώπη έχουμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση κατακεφαλή, δεκαπλάσια, σε σχέση με άλλα κρατημέλη όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία. Υπάρχει δηλαδή περιθώριο αύξηση της κατανάλωσης του βοηού σε πολλά κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε βεβαίως να, να μην περιμένουμε να υπάρχει και κάποια επίπτωση από την απότομη αύξηση της τιμής στο κύριο και της κατάστασης που προέκυψε στην Κίνα, αλλά ελπίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει προς όφελος των κτηνοτρόφων μας που παράγουν βόλιο. Και σε γενικές γραμμές θα πρέπει να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι δικοί μας οι καταναλωτές δεν ξεχνούν ότι το βόλιο είναι υψηλής αξίας θρεπτικό και αηφόρο προϊόν Κάτι που θα πρέπει να προβληθεί και στο μέλλον. Και τώρα να στραφώ και στους συναδέλφους μου που μπορούν να μιλήσουν για τις πτυχές του ανταγωνισμού. Ο Φλάβιο θα μιλήσει για τα θέματα του ε, εμπορίου. Ευχαριστώ Μάικλ. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντα τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Θα σα παρουσιάσω τη σκέψη μα ό,τι αφορά την πολιτική ανταγωνισμού στον τομέα τη γεωργία και κτηνοτροφία. Όπω ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και καιρό ασχολείται με τα θέματα του βοηού κρέατο, τη αγορά βοηού κρέατο και ιδιαίτερα την Ιρλανδική αγορά. Παρακολουθούμε τις πρόσφατες εξελίξεις όπως και εσείς και έχουμε τακτικές επαφές με τις αθηνικές αρχές ανταγωνισμού στην Ιρλανδία και όπως και η εθνικές αρχές ανταγωνισμού στην Ιρλανδία και εμείς είμαστε ανοιχτοί και πρόθυμοι για οποιαδήποτε συζήτηση και περιμένουμε στοιχεία ή τεκμήρια ή δεδομένα για να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους και να βελτιώσουμε την κατάστασή τους. Έχουμε δηλαδή κοινό στόχο μαζί, μαζί εμείς, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μάλιστα δεν θα πρέπει να γίνεται προσδιορισμός ε, τιμών σε κανένα επίπεδο της ε, της αλυσίδας, ε, ούτε από τους μεταπίτες ε, ε, τον, του κρέατος, ούτε από μεμονωμένους κτηνοτρόφους. Σε αυτό συμφωνούμε με τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού της, Ευρωπαϊ... της Ιρλανδίας. Όπως ξέρετε, το ενωσιακό δίκαιο επιτρέπει σε μεμονωμένους κτηνοτρόφους να οργανωθούν σε οργανώσεις παραγωγών και μέσω αυτών των οργανώσεων παραγωγών ε, οι κτηνοτρόφοι μπορούν από κοινού να προσδιορίσουν τις τιμές τους. Οπότε έχουν οι παραγωγοί τη δυνατότητα να προσδιορίσουν, συλλογικά όμως, τις τιμές των προϊόντων τους. Αρκεί να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις ε, που θεσπίζονται από το Ενωσιακό Δίκαιο. Ένα τέτοιο προπετούμενο είναι αυτές οι κοινά προσδιορισμένες τιμές να εφαρμόζονται στην παραγωγή βοήου κρέατος που η οργάνωση παραγωγών προσδιορίζει εκ μέρους των ε, όχι αυτό που αποφασίζουν δηλαδή μεμονωμένα η παραγωγή κτηνοτρόφη. Και το δεύτερο προαπαιτούμενο, η δεύτερη προϋπόθεση είναι η οργάνωση παραγωγών να ασκεί τουλάχιστον μία άλλη δραστηριότητα, συλλογικά δηλαδή, συλλογική δραστηριότητα προ όφελο, προ το συμφέρον των παραγωγών. Δηλαδή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο τέτοιε δραστηριότητε. Και αυτό αφορά την προμήθεια, ε, συσκευασία, σήμανση, έλεγχο, ποιότητας και ούτω καθεξής. Πάντως, μάθαμε ότι στην Ελλανδία ήδη αναγνωρίστηκαν το Σεπτέμβριο οι πρώτες δύο τέτοιες ε, οργανώσεις παραγωγών, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, πολύ πρόσφατα δηλαδή έγινε αυτή η διαπίστευση, η αναγνώριση. Δεν υπάρχουν όρια για το μέγεθος του, της οργάνωσης παραγωγών. Θα μπορούσαν και όλοι οι αγρότες της Ιρλανδίας να προσχωρήσουν ε, σε μία ή δύο το πολύ οργανώσει παραγωγών. Οπότε αυτή είναι η τάση. Το ενωσιακό δίκαιο προβλέπει μηχανισμού για να γίνει συλλογικό προσδιορισμό των τιμών από του παραγωγού, προκειμένου να αντισταθμιστεί η αγοραστική δύναμη των μεταποιητών του κρέατο. Και νομίζω ότι είναι δίκαιε αυτέ οι εξέλιξει, γιατί θεωρούμε ότι οι οργανώσει παραγωγών είναι ο μόνο βιώσιμο ε, φορέα για την προάσπιση των συμφερόντων των κτηνοτρόφων. Δεν ε, βρισκόμαστε εμεί απομονωμένοι ε, στις Βρυξέλλες έναν ε, χρυσελεφάντινο πύργο και τα βλέπουμε αφιψηλού. Μάλιστα είχαμε μία μελέτη το Μάιο του 2018 που δημοσιεύθηκε και ήταν μία πολύ εμβριθής μελέτη ε, για τις οργανώσεις παραγωγών και εκεί αναφέρεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών ασκούν συλλογικά είτε σε αναγνωρισμένη είτε σε άτυπη οργάνωση να προσδιορίσουν όχι μόνο τις τιμές, αλλά και να ασχοληθούν και με άλλες δραστηριότητες που ενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους. Για παράδειγμα, φαίνονται από στατιστικά στοιχεία, γιατί αυτή η μελέτη κάλυπτε το τομέα βοήου κρέατος. Εκεί πάνω από το 90% των ε, οργανώσεων που ερωτήθηκαν ε, μίλησαν για κοινέ στρατηγικέ ε, εμπορευματοποίησει, συμβάσει, ποσότητα και ποιότητα και δύο τρίτα των οργανώσεων παραγωγών ε, δήλωσαν ότι έχουν και άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης αποτελεσματικότητας τη αποτελεσματικότητά στα κράτη-μέλη. Και οι τρει άλλε δραστηριότητε που εφαρμόζονταν πιο συχνά ήταν η έλεγχη ποιότητα, η συγκέντρωση προϊόντων και διανομή και μεταφορά. 92% των ε, φορέων που ερωτήθηκαν ασκούσαν και τουλάχιστον μία ακόμη δραστηριότητα από το από την απαιτούμενη μία δραστηριότητα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και 69% τέτοιων οργανώσεων είχαν και δύο, τρεις τέτοιες παρόμοιες δραστηριότητες ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και όχι μόνο την ε, απαιτούμενη από τον νόμο μία τουλάχιστον. Οπότε μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ε, το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που θεωρούν ότι προέρχεται από την οργάνωση παραγωγή είναι η σταθερότητα των τιμών, η δημιουργία οικονομιών κλίμακος, η βελτίωση του βιωτικού του επίπεδου και η βελτιωμένη πρόσβασή τους στην αγορά. Οπότε μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους κτηνοτρόφους ε, να οργανωθούν σε οργανώσεις παραγωγών, γιατί αυτός είναι ο τρόπος να αποφύγουν ε, προβλήματα με το δίκαιο ανταγωνισμού. Και μάλιστα έχουμε ήδη απτές αποδείξεις ότι έχουν γίνει τα πρώτα βήματα και σε άλλους τομείς και είναι πραγματικά εργαλείο αλληλοβοήθειας μεταξύ των παραγωγών η δυνατότητα οργάνωσης τους σε οργανώσεις παραγωγών. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε απορίες σας στη συνέχεια. Και πριν περάσουμε στη συζήτηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο και στο συνάδελφο από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ευχαριστώ. Ε, θα επικεντρωθώ ε, στο ερώτημα γιατί θεωρείται το προϊόν το βόλιο κρέας ε, στο εμπόριο. Υπάρχουν κάποιες διαρθρωτικές αδυναμίες του ίδιου του κλάδου, ακούσαμε και προηγουμένως τα στοιχεία και αυτό αντανακλά ε, και στις διαπραγματεύσεις και είναι δύσκολο βέβαια να απομονώσουμε το βόλιο κρέας από τα άλλα στοιχεία των διαπραγματεύσεων για τη γεωργία, γενικότερα των διαπραγματεύσεων για τις εμπορικές συμφωνίες. Είναι σημαντικό όμως σήμερα εδώ να επικεντρωθούμε στην ιδιαιτερότητα του βοηού κρέατος που είναι ευαίσθητο προϊόν και το ξέρουμε σε όλες τις διαπραγματεύσεις με τους ανταγωνιστές μας, προμηθευτές βοήου. Και στην ουσία αυτό ε, έχει αντανάκλαση, αλλά και στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Γιατί τα πιο ευαίσθητα προϊόντα εξαιρούνται από τις αρχικές συμφωνίες και ε, υποχωρήσεις και πάνε προς το τέλος της συμφωνίας. Επίσης, ε, σταθμίζονται πάρα πολύ προσεκτικά ε, με μελέτες αντικτύπου, με ε, περιστατωμένη και σχολαστική εξέταση των συνθήκων που επικρατούν στην αγορά και έτσι ώστε να ανοίγουμε τις αγορές μας με τρόπο που να έχει νόημα για τους εταίρους με τους οποίους διαπραγματευόμαστε, αλλά να μας επιτρέπουν να υπερασπιζόμαστε και να προασπίζουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων κτηνοτρόφων. Αυτή η ιστορία λοιπόν με το βόιο ε, κρέας ακολουθήθηκε σε όλες τις διαπραγματεύσεις στη ΣΕΤΑ. 20.000 ε, τόνοι για το 2019 είναι το βόηο κρέας που επιτρέπεται. Ωστόσο, οι εισαγωγές βοηού κρέατος ε, από τον Καναδά είναι ε, 600.000 τόνοι ε, ε, σε σφάγια. Ε, είναι το 3% περίπου. Δεν νομίζω ότι ο Καναδάς μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι παραπάνω από ένα πολύ μικρό κλάσμα της ποσόσης, γιατί είναι πάρα πολύ δαπανηρό να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή γραμμή παραγωγής χωρίς ορμόνες για εξαγωγή στην Ευρώπη. Δεν είναι ανταγωνιστικό αυτό ε, οπότε δεν έχουν καλύψει την ποσόστοση. Μερκοσούρ, που είναι φυσικά το μεγάλο ερωτηματικό εκεί που έχετε πολλοί από εσά. Ε, συμφωνήσαμε με τις χώρες Μερκοσούρ, 99.000 τόνους, μια ποσόστοση ε, που σταδιακά θα μπει σε έξι ίσα βήματα μέσα σε μια πενταετία. Αυτό το βλέπουμε στο γενικό πλαίσιο, γιατί ήδη εξάγουν οι χώρε Μερκοσούρ προ την Ευρώπη 200.000 τόνου ετησίω περίπου βοήου. Για 50-60.000 τόνου περίπου αυτής της ποσότητας ε, πληρώνονται πλήρη δεσδασμή, εκτός ποσόστοσης. Και η πρώτη συνέπεια, πιστεύουμε, της ποσόστοσης θα είναι εξής. Εκτός από αυτές τις εισαγωγές, εκτός ποσόστοσης, μάλλον ένα τμήμα θα ενταχθεί ε, στην ποσόστοση των 99.000 τόνων. Δηλαδή δεν θα έχει όλη η ποσότητα ε, επίπτωση στην αγορά. Εκτός αυτού υπήρξε και ένας κατακαιρματισμός. 55% ε, αφορά τον οπό ε, βόιο κρέας που είναι και το πιο ευαίσθητο προϊόν γιατί είναι και τα τεμάχια που είναι της καλύτερης ποιότητας και τα πιο ακριβά και το 45% που είναι λιγότερο ευαίσθητο αφορά το κατεψυγμένο βόλιο κρέας. Φυσικά ε, αυτά τα ποσοστά θα πρέπει να τα δούμε στο πλαίσιο ε, της ε, κατανάλωσης και παραγωγής στην Ένωση που είναι περίπου 8 εκατομμύρια τόνοι το 2018 είναι λίγο παραπάνω από το 1% αυτή η ποσόστοση από Μερκοσούρ της κατανάλωσης στην Ένωση. Και εκτός αυτού, αν υπάρχουν οποιασδήποτε ανησυχίες για τον αντίκτυπο, υπάρχει μια ασφαλιστική κλίδα διμερής που μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν αυξάνονται οι εισαγωγές ή όταν ε, υπάρχει πραγματική στρέβλωση της αγοράς ή προβλήματα. Γιατί τα λέω αυτά. Ε, διότι το προϊόν αυτό είναι ευαίσθητο, είχε την αντίστοιχη μεταχείριση και έχουν αναλυφθεί δεσμεύσεις ε, που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη δυνατότητα της αγοράς να απορροφά τις συγκεκριμένες ποσότητες. Από την άλλη, ε, είναι γεγονός ότι το βόηο είναι ευαίσθητο και για τους εταίρους μας ορισμένους, το είπαν και οι συνάδελφοι, υπάρχουν εξαγωγές της Ένωσης που παίζουν σημαντικό ρόλο και νομίζω θα εξακολουθήσουν στο μέλλον ε, να παίζουν ένα ακόμα σημαντικότερο ρόλο. Έχουμε πλεόνασμα στα προϊόντα βορείου κρέατος, 500.000 τόνους σε ε, εξαγωγές ετησίως. 160.000 είναι πλεονασματική. Εδώ λαμβάνει την υπόψη και το βόηο κρέας. Ε, ε, αν βάλουμε μάλλον και το βόηο και τα ζώντα ζώα, το πλεόνασμα φτάνει στις 400.000 τόνους. Ε, οπότε είναι για την παραγωγή μας οι εξαγωγές πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε συμφωνίες προτιμησιακές με χώρες που απορροφούν μεγάλο τμήμα αυτών των εξαγωγών, όπως είναι η Τουρκία, Βοσνία, Ισραήλ, Ελβετία και άλλες. Ε, είναι προτιμησιακοί εταίρη μας. με το ειδικό προτιμησιακό καθεστώς. και βλέπουμε το εμπόριο να μην εμποδίζεται ή να μην διαστρεβλώνεται από ε, περιτά υγειονομικά μέτρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το προϊόν, το εξαγωγικό. Και στο μέλλον περιμένουμε να αυξηθούν οι ευκαιρίε και οι δυνατότητε. Όταν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία με το Βιετνάμ, θα απελευθερωθεί το βόλιο μετά από τρία χρόνια. Είναι πολύ ελπίδοφόρα η αγορά. Και με την Ιαπωνία επίση σιγά σιγά εγκαταλείπεται η εξαγωγή των ζώων των ζώων. έχουμε όμως σταδιακή αντικατάσταση από μία ποσόστοση για το κρέας. Άλλες ε, προβλέψεις και... Να τελειώνετε σιγά σιγά παρακαλώ λέει ο πρόεδρος αν γίνεται. Ναι, ολοκληρώνω. 20 λεπτά δεν είχα. Έφτασα στα 20 λεπτά. Όχι, είχατε 20 λεπτά συνολικά. Ε, είναι πολύ ευνοϊκέ οι εξελίξει λοιπόν σε ό,τι αφορά τη ζήτηση και τη εγχώρια αγορά και τη εξαγωγική. Ε, η εγχώρια αγορά παραμένει ε, βέβαια οι βασικότεροι, αλλά έχουμε τις αναδυόμενες οικονομίες και χώρες που αρχίζουν να ζητούν ε, στην Ασία και στην Αφρική όσο αναπτύσσεται η αστική τους και η μεσαία τάξη και ελπίζουμε να ε, αυξηθούν οι εξαγωγές μας προς τα εκεί. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν, ε, ακριβώς για να υποφεληθούμε από αυτές τις εξαγωγικές ευκαιρίες, όπως είπα προηγουμένως και ιδιαίτερα για την Κίνα που είναι το υπαριθμόν ένα κράτος μαζί με το Χονγκ Κόνγκ, η εξαγωγική αγορά, ε, καλό είναι λοιπόν να αξιοποιήσουμε πλήρως, να υποφεληθούμε και να περάσουμε πέρα από τα εμπόδια που έχουμε ήδη από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Πέντε είναι τα κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή εξάγουν στην Κίνα. Αλλά είμαστε πολύ ε, ε, δεσμευμένοι με αυτές τις χώρες. Περιμένουν και άλλες επτά, θέλουμε και άλλες χώρες να αυξηθούν και πιέζουμε πολύ την Κίνα να καλυφθεί ε, το έλλειμμα πρωτεΐνων που έχει προκληθεί από την Αφρικανική Πανόλη του Χείρου και να μπορέσουμε να εξαγάγουμε σε αυτή τη τεράστια αγορά. Ευχαριστώ πολύ ε, τους τρεις εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις παρουσιάσεις αυτές. Διαπιστώνω ότι οι συνάδελφοι έχουν πολύ μεγαλύτερη πειθαρχία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την τήρηση του χρόνου αγόρευσης. Εν πάση περιπτώσει, ας έρθουμε τώρα στις ερωτήσεις. Ήδη έχω ε, μερικούς συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Σημειώνει ονόματα η γραμματεία. Η κυρία Μαγκίνες πρώτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μήπως η κυρία Σαντέρ προηγητώ γιατί έχει μια συνάντηση μετά και ευχαρίστω παραχωρώ τη θέση μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Όντως, θα ήθελα να κάνω μια σειρά από ερωτήσεις με τη σειρά μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πρώτα απ' όλα το τομέας της Ευρώπης για το βόλιο κρέας είναι καθοριστική σημασία για την κοινοτροφία μας είναι ευπαθής τομέας και γνωρίζει σήμερα ιδιαίτερες πιέσεις. Έχουμε λοιπόν προβλέψει και σκεφτεί μια σειρά από ιδέες για μια στρατηγική προσέγγιση που θα επέτρεπαν να ε, ενισχύσουμε αυτόν τον τομέα. Χάρη στην γεωργική πολιτική του 2013 και τη μεταρρύθμισή της, στα πλαίσια της πρότασης Omnibus το 2018, διαθέτουμε ήδη μια σειρά από ε, ενισχυμένα εργαλεία ω προς τις οργανώσει, την ε, κατανομή των συμβάσεων, την συλλογική διαχείριση κινδύνων και ούτω καθεξής. Πρώτη μου ερώτηση λοιπόν πώς έχει πάει η υλοποίηση του συνόλου των εργαλείων αυτών για τον τομέα της κτηνοτροφίας που παράγει βόλιο και μετά για την τρέχουσα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Έχουμε δύο επιπλέον εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν με οικονομική υποστήριξη. Τα επιχειρησιακά προγράμματα και τα, οικο, τα οικολογικά συστήματα. Πώς να ανταποκριθούμε λοιπόν μέσω αυτών στι μελλοντικέ προκλήσει. Λυπάμαι, αλλά δεν θα μείνω για να ακούσω τι απαντήσει, θα μου τα πούνε οι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μακίνα τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση. Τρει ερωτήσει θέλω να θέσω προ του τρει συναδέλφου τη Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα για την DG Competition. Είχαμε προηγουμένω μια συζήτηση στο περιθώριο. Θα μπορούσε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να πει ότι δεν υπάρχουν πρακτικέ που να παραβιάζουν του κανόνε ανταγωνισμού στον τομέα παραγωγή βοήου. Και τι γίνεται με τη συνδεδεμένη βοήθεια, όπου έτσι και αλλιώ όλα τα προϊόντα κρέατο έχουν την ίδια προσφορά ω προ την τιμή στην αγορά. Πώ το βλέπει αυτό η αρχή ανταγωνισμού στην ε, DG για, την τον ανταγωνισμό, τι θα κάνετε για τι πρακτικέ που παραβιάζουν αυτού του κανόνε. Και ευτυχώ αυτοί, αυτές οι... οι δύο φορέ ιδρύθηκαν στην Ιρλανδία για τον κύριο Σκάνελ. Ε, είπατε πώ άλλαξε η κατηγοριοποίηση, το πώ διαθέτονται στι διάφορε κατηγορίε τα προϊόντα κρέατο. Ε, μπορείτε να πείτε περισσότερε λεπτομέρειε και για τι εισαγωγέ από την Νότιο Αμερική. Ε, καταλαβαίνω ότι τρώμε πολλέ μπριζόλε και αυτό έχει επίπτωση και στην αγορά. Ε, μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Η συνάδελφος Αγγιλάρ. Είναι προφανές και το σχολιάσαμε ήδη, ότι ο ευρωπαϊκό τομέα βόλου κρέατο είναι αυτό που επηρεάζεται κυρίω από τον Brexit. Και οι εμπορικέ συμφωνίε Ευρωπαϊκή Ένωση που διευκολύνουν την εισαγωγή φθηνού κρέατο ε, χαμηλότερη όμω ποιότητα από το δικό μα και οι χαμηλέ τιμέ οδηγούν του κτηνοτρόφου μα να πολλούν μερικέ φορέ σε τιμή κάτω του κόστου παραγωγή. Και στην πατρίδα μου την Ισπανία Έχουμε 3,4 δις ε, τζίρο το χρόνο και 150.000 οικογένειες που βιοπορίζονται από τον τομέα αυτό και ιδιαίτερα για το βόλιο θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε τεράστια γραφειοκρατία λόγω της ΚΑΠ για τους ε, κτηνοτρόφους βόλιο κρέατος και μάλιστα γίνεται μια εκστρατεία ε, κυλίδωσης του ευρωπαϊκού κτηνοτροφικού κλάδου και είναι το θύμα αυτής της συκοφαντικής εκστρατείας ο τομέας αυτός. Θέλουμε λοιπόν περισσότερη προβολή και νέο σύστημα επισήμασης ε, του κρέατος. Θέλουμε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση στην κατανάλωση, τις νέες τάσεις και για τις επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών ε, μέχρι το 2025. Επίσης, συμφωνίες με τη Νέα Ισλανδία και την Αυστραλία ίσως επηρεάσουν αρνητικά τον τομέα βοιοκράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να το σχολιάσετε. Ευχαριστώ κύριο Σκαλινόφσκι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, τι απειλές θα έχουμε στο μέλλον για τον τομέα βοήου κρέατος από την Νέα Πράσινη Συμφωνία. Επίσης, στην Πολωνία, όπως είπατε, ε, είναι ε, σε δραματικά χαμηλά επίπεδα οι τιμές βοήου κρέατος. Και ο περιορισμός ε, των πολωνικών πωλήσεων βόλιο κρέατος στην Τουρκία επιδίνωσε την κατάσταση. Το 2018 η Πολωνία εξήγε πάνω από 33.000 ε, τόνους ε, νοπού βόλου κρέατος. Το 90% του συνολικών ευρωπαϊκών εξαγωγών δηλαδή προς την Τουρκία. Ενώ τον Ιούλιο και Αύγουστο είχαμε απόλυτη κατάρρευση της αγοράς. Και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προετοίμασε ε, αντισταθμιστικό πακέτο για την αποζημίωση των ε, κτηνοτρόφων. Ενώ είναι αδύνατο να μην ερμηνευτεί αυτή η απροθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το στηρίξει ως άνηση μεταχείριση. Γιατί λοιπόν δεν ετοίμασε τέτοιο πακέτο στήριξης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Άλιμοφ. Ευχαριστώ. είναι Обединеното кралство и Ирландия са лидери в говеждо. Ε, ο τομέας του βοηού κρέατο στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένο. Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι ε, πρωτοπόροι ε, στην παραγωγή βοηού κρέατο. Οι χώρε όμω της Ανατολική Ευρώπη καλύπτουν τις ανάγκες τους κυρίως μέσω των εισαγωγών. Και οι κτηνοτρόφοι εκεί κερδίζουν κάτι ψίχουλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους στηρίξουμε. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται οπωσδήποτε αυτή τη στήριξη οικονομική. Εάν θέλουμε να αποκλείσουμε τους κτηνοτρόφους μας από αυτή την οικονομική βοήθεια, αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά και θα απειλεί στην ανάπτυξη της υπαίθρου την ίδια. Ερωτώ λοιπόν τι προτίθεται να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος. Μέχρι τώρα είχαμε συνδεδεμένες ενισχύσεις και κρατικές ενισχύσεις. Η κυρία Σμιτ Μπάουερ. Όπως ακούσαμε σήμερα, έχουμε 4,5% μείωση το τελευταίο διάστημα. Ανησυχούμε και το Brexit και το Mercosur. Είναι αύριο. Έχουμε και την κλιματική αλλαγή και ακραία καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν ε, και τις ζωοτροφές και η μείωση της κατανάλωσης είναι για μας μεγάλη πρόκληση. Κατά τη δική μου άποψη, οι επιπτώσεις στην αγορά βοηού κρέατος στο Mercosur ε, στην αντίστοιχη έκθεση αντικτύπου δεν αντανακλώνται και δεν αναλύονται με τρόπο ρεαλιστικό, ε, διότι γίνεται λόγος ε, για εισαγωγές, αλλά δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα στην ποιότητα. Έχουμε τα πιο ευγενή τεμάχια που έχουν άλλη τιμή. Ε, δύο είναι τα θεωρητικά σενάρια στα οποία βασίζεται η μελέτη αντικτύπου. Για ποιο λόγο όμως δεν βασίζεται ε, στο πραγματικό, υπαρκτό, σημερινό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Γιατί δεν κάνατε με βάση αυτά τη μελέτη. Και επίσης ε, έχω αναφερθεί σε μελέτες ειδικέ αναχώρα για τις επιπτώσεις. Και επίσης Ωραίο είναι το πακέτο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για βοήθεια, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ευχαριστώ η κυρία Κατάινεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι η παγκοσμιοποίηση παίζει όλο ένα και μεγαλύτερο ρόλο στην αγορά παραγωγής και στην παραγωγή τροφίμων. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε τρόφιμα καλύτερης ποιότητας ε, και να είμαστε βέβαιοι ότι τέτοια παράγονται και θα πρέπει να προστατεύουμε τη διατροφική αλυσίδα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι ε, και ενημέρωση ακόμα και για τα σούπερ μάρκετ ε, όπου καταλήγουν τα προϊόντα να διατίθενται στη διατροφική αλυσίδα. Θα πρέπει οι προϋποθέσεις του εισαγόμενου, που ισχύουν και το εισαγόμενο κρέας είναι οι ίδιες όπως για το ευρωπαϊκό. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχουμε κανόνες αυστηρούς προέλευσης για κρέας από τη Λατινική Αμερική, από την Αργεντινή, από την Αργεντινή ας πούμε. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Τεσέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο τομέας της κτηνοτροφίας και ειδικά οι κτηνοτρόφοι βόηου αντιμετωπίζουν δυσκολίες είναι για τα τελευταία χρόνια αυτός ο κλάδος επένδυσε πολλά για να βελτιώσει τις συνθήκες παραγωγής και ως προς τη ζωική ευζοία και ως προς τα περιβαλλοντικά και οικολογικά μέτρα. Τον τομέα αυτό λοιπόν τον φέρνουμε να ανταγωνιστεί χώρες όπου οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις παραγωγής δεν είναι καθόλου οι ίδιες. Δείτε τι συμβαίνει με τις χώρες του Μερκοσούρ. Ο αριθμός ζώων που, που εκτρέφονται ως προς την επιφάνεια μιας εκμετάλλευσης είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τους αυστηρούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον αριθμό ζώων που επιτρέπονται αναεκτροφείο. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Πώς θα τα λάβουμε αυτά υπόψη την, τις προποθέσεις εντός των οποίων ζουν τα ζώα στο επίπεδο των εμπορικών μας διαπραγματεύσεων, δηλαδή πέραν της ποσότητας κρέατος, των τόνων που εισάγουμε, πρέπει να μας απασχολήσει και η ποιότητα. Πρέπει μάλιστα να επαγρυπνούμε και να λαμβάνουμε υπόψη και τις απαιτήσει του καταναλωτών ως προς αυτό. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ρίτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με κάλυψαν σε ορισμένα σημεία οι συνάδελφοι. Έχουμε, είχαμε πραγματική ε, μείωση της ε, των τιμών βοηδού κρέατος που δημιούργησε τεράστια, ε, τεράστια ένταση μεταξύ των κτηνοτρόφων και της, των υπόλοιπων κρίκων τη αλυσίδα. Δυστυχώ ήταν αδιαφανής ε, η αγορά βοηθού κρέατο και δεν υπήρχαν συνθήκε θεμητού ανταγωνισμού και λόγω αυτή τη έλλειψη ανταγωνισμού και τη αδιαφάνεια ε, έχουμε μείωση και τη ποσότητα τη διακίνηση των προϊόντων θεωρείτε ότι είναι δίκαιο το μερίδιο της τιμής που λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι ή όχι. Και σε σχέση με αυτά που είπαν η κυρία Γκυλάρ και ο κύριος Δεσέρλ, ήδη αναφερθήκαμε στο ζήτημα των ε, εισαγωγών που ρίχνουν τις τιμές του κρέατος. Εγώ έχω μια διαφορετική ε, εντύπωση. Θεωρείτε ότι είναι λάθος να περιμένουμε από ε, τις, τους παραγούς των τρίτων χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου να πληρούν τις υψηλές ε, ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τρόφιμα για το περιβάλλον. Έχει νόημα να εισάγουμε τρόφιμα που δεν έχουν τα ίδια πρότυπα και τις προδιαγραφές με τα δικά μας. Ο κύριος Ντάβιτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη ε, με κάλυψαν οι προλαλήσαντες για κάποιες ερωτήσεις. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση για τη δική μου την πατρίδα, την Τσεχία. Ε, τα τελευταία 30 χρόνια είχαμε μείωση της ε, ε χώρας παραγωγής κατά το ίμιση, γιατί είναι πολύ φθηνές τιμές του βόηου κρέατος και οι εξαγωγές ε, κατευθύνονται κυρίως προς τα Βαλκάνια, τις Βαλκανικές χώρες και την Τουρκία. Τώρα αναμένουμε να μειωθούν οι μεταφορές ζών των ζώων σε μεγάλες αποστάσεις. Οπότε θα έχουμε τεράστιες ε, ε, ζημιέ στον κλάδο. Πώ θα τι αντισταθμίσουμε, πώ θα αποζημιώσουμε του κτηνοτρόφου, Η κυρία Πύρικ. Πρόεδρε, έγιναν ήδη πολλέ ερωτήσει. Εγώ έχω μια ερώτηση για το ψήφισμά μα για την Τουρκία που περάσαμε πριν από δύο εβδομάδε στο Στρασβούργο. Εκεί γίνεται λόγο για κυρώσει εξαγωγικέ από την Τουρκία στην Ευρώπη, εισαγωγίες για την Ευρώπη. Αλλά τι θα γίνει εάν η, η Τουρκία σταματήσει τις εισαγωγές ε, που μπορεί να μην είναι υψηλές, αλλά είναι βόλιο κρέας. Ε, και τι ε, ε θα γίνει, ε, έχετε προβλέψει αποζημιώσει για τους αγρότες, γιατί είχαμε και το προηγούμενο της Ρωσίας με τα αντίπεινα ε, ως προς τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων. Ευχαριστώ, κύριος Λεμπρετών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το βόλιο κρέα είναι προϊόν ευαίσθητο γεγονό. Στη Γαλλία χάσαμε ε, ένα εκατομμύριο ζώα σε τρία χρόνια. Ε, από 19,5 ε, εκατομμύρια σε 18,5. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Δεν άκουσα πολλές λύσεις. Εξού και η πρώτη μου ερώτηση. Αντί ε, να γκρινιάζουμε για τις μικρές εκμεταλλεύσεις, δεν θα πρέπει να έχουμε μια θελησιοκρατία με ενίσχυση των τιμών και εξυγχρονισμό και με βοήθεια των εκμεταλλεύσεων. Και μήπως θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε καλύτερα τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών για να αποφεύγουμε την εισαγωγή βοηού. Μιλήσαμε για το ΣΕΤΑ. Τώρα θα κάνει μεγάλη ζημιά και το και θα έχουμε και συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να έρθουν 35.000 τόνοι. Είναι ε, μεταβλητή προσαρμογή στο κόστος στο βόλιο κρέα. και σε ποια αριθμητικά στοιχεία βασίζεται η Επιτροπή για να δίνει ποσοστό βοήου κρέατος σε τρίτες χώρες. Ευχαριστώ κύριο Φλάναγκα. Ε, Ευχαριστώ για αυτή τη διαφωτιστική συζήτηση Απλώς θέλω να καλωσορίσω τους παραγωγούς του Galway από την βορειοδυτική Ιρλανδία για να ακούσουν και εκείνοι τι συμβαίνει εδώ. Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Σκάνελ από την Επιτροπή για την κατεπίγουσα κατάσταση στον τομέα του Βόλου και τα μέτρα βοήθειας. Ο κανονισμός που εγκρίθηκε για να επιτρέψει να εκταμιευτούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ για να αποζημιωθεί η Ιρλανδία προέβλεπαν δημοπρασίες για να δούμε αν οι θέλουν να μειώσουν το κόστος παραγωγής ή κατά πόσο μπορούσαν να θέσουν συγκεκριμένους στόχους όπως με οικολογικά προγράμματα, προγράμματα διαφοροποίησης, βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων και της αηφορία των εκμεταλλεύσεων. Εδώ λοιπόν, προτού αυτό περάσει, ήθελα να εκφράσω τις έντονες ανησυχίες μου ως προς την κοινότητα των κτηνοτρόφων. Οι δημοπρασίες αυτές δεν θα γίνουν στην πραγματικότητα και μόνο ένα πράγμα θα εφαρμοστεί. Μείωση του κόστους παραγωγής. Ε, θα μου πείτε ίσως ότι αυτό δεν θα συμβεί εσείς, αλλά πραγματικότητα είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Λίνσεν, ο υπεύθυνο του Υπουργείου για τα θέματα κτηνοτροφίας, είπαν στην Αρμόδια Επιτροπή ότι δεν υπάρχει κανένας πληστηριασμός υπόψη, καμιά δημοπρασία. Το μόνο που θα γίνει είναι η μείωση του κόστος παραγωγής σας. Έγραψα και στο γραφείο σας, εξηγώντα τη συγκεκριμένη περίπτωση και φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει αυτή η επιλογή για την Ιρλανδία γιατί λοιπόν έγινε αυτό και γιατί οι πλέον αηφόροι παραγωγοί βοιού στον κόσμο, οι Ιρλανδοί, ε, έχουν αυτή την απέτηση απέναντί τους να μειώσουν το κόστος τη παραγωγής, ενώ έχουμε 19 τόνους βόηου από χώρε που χρειάζεται να κάψουν τροπικά δάση για να παράγουν το βόηο. Ευχαριστώ κύριο Κούσμιουκ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις τρεις γενικές διευθύνσεις για την παρουσίαση που μας έκαναν. Βέβαια, μας παρουσίασαν μια πιο αισιόδοξη θεώρηση της αγοράς του βοηού κρέατος. Ενώ βλέπουμε ότι οι τιμές του βοηού κρέατος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, αλλά και σε μεμονωμένες χώρε όπω την Πολωνία, είναι χαμηλές που και δεν δικαιολογούν τέτοια αισιοδοξία. Έχω μία ερώτηση τι θα γίνει στο μέλλον με το Βόλιο Κρέα αν ολοκληρωθεί η υπογραφή της συμφωνίας με τις χώρες Μερκοσούρ δεδομένου ότι από τις τέσσερις χώρες αυτές θα έχουμε το 70% των εισαγωγών, του συνόλου των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε και στο μέλλον στους αυξηθούν αυτές οι εισαγωγές. Ενώ γνωρίζουμε ότι οι παραγωγοί αυτών των χωρών δεν πληρούν τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές που ισχύουν για τους Ευρωπαίους γεωργούς. Οπότε εγώ Βλέπω μόνο απεισιοδοξία και επιδείνωση της κατάστασης από τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας με το Μερκοσούρ. Ευχαριστώ. Κύριος Μπούντα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε τι τεράστιες ε, θυσίες κάνουν οι Μας είπατε ότι δεν τους μένει παρά να οργανωθούν. Μας είπατε ότι δεν μένετε απομονωμένοι σε ένα ξελεφάντινο πύργο, αλλά έχετε επαφή με την πραγματικότητα. Γνωρίζετε όμως ότι αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία ε, ένα κιλό ε, κρέας βόηο κρέας στη 1,5 ευρώ, ενώ το κόστος παραγωγής είναι πάνω από 2 ευρώ. Μήπως λοιπόν θα οδηγηθούμε σε εξαφάνιση της εκτροφής ε, βοηδών. Γιατί αν ε, η τιμή πώληση είναι χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής, θα αναγκαστούν να κλείσουν τις κτηνοτροφικές τους μονάδες οι κτηνοτρόφοι μας. Επίσης, τι γίνεται με τις εξαγωγές και εντός Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να δώσουμε κάποιες ευκαιρίες στους κτηνοτρόφους δεν μπορούμε να τους αφήνουμε στη μοίρα τους ενώ βρίσκονται στο χείλο της χρεοκοπίας και εμείς να εισάγουμε χειρότερης ποιότητας ε, κρέας από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας των εισαγόμενων κρεάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξεπλάγει όταν άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων στην Κίνα επηρεάζει την αγορά βοηοκρέατος. Αυτό δεν ευσταθεί. Αν μια χώρα δεν παράγει πια αρκετό κρέας, δεν μπορεί παρά, ε, χείριο, δεν μπορεί παρά να <clears throat> καταναλώνει περισσότερο βόιο. Επίση, Αφρικανική Πανόλη των Χείρων είχαμε και στην Ευρώπη. Πριν από πέντε χρόνια είχαμε στι χώρε τη Βαλτική, στην Πολωνία και σε άλλε οχτώ χώρε τώρα πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τέτοια κρούσματα και σε εμά. Τι επιπτώσει είχε η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ επηρέασε το τη δική μα αγοραβού κρέατο και πώ θα την επηρεάσει και στο μέλλον, στην επόμενη πενταετία. Στι Βαλτικέ χώρε παράγουμε μόνο το 50% του κρέατος που καταναλώνουμε, οπότε αναγκαζόμαστε να εισάγουμε το υπόλοιπο 50% χείριου κρέατος. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τι επιπτώσεις έχει ήδη ασκήσει η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων στον τομέα του βοήου κρέατος στην Ευρώπη τώρα, αλλά και τις συνέπειες που θα έχει την επόμενη πενταετία. Γιατί δεν έχουμε κάνει αρκετά για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Γκερέρο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω εδώ τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη, διότι όταν μιλάμε για εξαγωγές και εμπόριο του βόηου, χωρίς και τις άλλες κατηγορίες του κρέατος, δεν γίνεται να βγάλουμε νόημα για τις επιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας είπαν τι γίνεται με την αύξηση ε, των εξαγωγών, ιδίως προς χώρες που υπάρχει πρόβλημα με την κατανάλωση. Το είδαμε με τα όσα συμβαίνουν στην Κίνα και τι σχετικέ εξαγωγέ. Η αύξηση των εξαγωγών θα έχουν επιπτώσει όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά παγκοσμίω. Και το πρόγραμμα που μα ε, υποβάλλατε θα έχει, σημαντική, σημασία, θα έχει μεγάλη σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Μετά για τη Γενική Διεύθυνση Trade, σίγουρα χρειάζονται φιλοδοξότερε προτάσει για να βελτιώσουμε του κανονισμού και την εξαγωγή ζών των ζώων, ιδίω για χώρε εκτό Ευρώπη, που αναφέρθηκαν ήδη, όπω η Τουρκία και το Ισραήλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γιούγκε. Ευχαριστώ. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας ανέφεραν ε, τα αίτια που οδήγησαν στην κρίση στο κρέας και πρότειναν ε, κάποιες λύσεις, ε, μεταφορές από τον πρώτο πυλώνα, προώθηση, καλύτερη προβολή των προϊόντων και κάποιες εμπορικές συμφωνίες. Παρ' όλα αυτά, οι χαμηλές τιμές κρέατος στην Πολωνία οφείλονται στις άνισες συνθήκες ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή αγορά και η Πολωνία έχει χαμηλότερες άμεσες ενισχύσεις. Βρίσκεται στο 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου το επίπεδο άμεσων ενισχύσεων στην Πολωνία. Οπότε έχετε αναλύσει την επιρροή της, ανι... της ανισότητας της άμεσης ενισχύσης μεταξύ των Ευρωπαίων παραγωγών. Μήπως και αυτές έχουν συμβάλει, αυτές οι διαφορετικές άμεσες ενισχύσεις, στην κρίση στην αγορά βιοκρέατος και μήπως θα έπρεπε να, να αποκαταστήσει το θεμητό ανταγωνισμό προωθώντας κάποιες ενέργειες για την ε, εξίσωση των συνθηκών. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δύο ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα για την κατανάλωση του κράτους στην Ευρώπη ως τελικατέσεν. Ε, πόσο καταναλώνονται τέτοια προϊόντα και ε, τι αύξηση προβλέπεται να υπάρχει. Και για το μέλλον και τον, του ανταγωνισμού. Τι επιπτώσεις θα έχει η παραγωγή σε επίπεδο εργαστηρίων, τεχνητού κρέατος, πειραματικός. Υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης μιας τέτοιας αγοράς. Για την ώρα πολλά φαίνεται να είναι έτοιμα, αλλά δεν είναι αντικείμενο εμπορίας. Η κυρία Βίνα, ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, να συνοψίσω, κατάλαβα καλά ότι τα αίτια αυτής της κρίσης έχουν να κάνουν με την ε, υπερπαραγωγή ε, με αδιαφάνεια και με ποιότητα, με ανισότητες και αδικίες που δεν μπορούμε να αντιτρήσουμε. Γι' αυτό πέφτουν οι τιμές. Για ταυτόχρονα η, η παραγωγή μας πρέπει να παράγουν κάτω του κόστους γιατί έχουν το ανταγωνισμό από χώρε με παραγωγή που είναι πιο φτηνή. Εκεί παράγεται. Δεν ακούσαμε σήμερα το πρωί για τη μεγάλη μελέτη που όλα τα σενάρια του μέλλοντος εξακολουθούν να πιέζουν τους μικρούς αγρότες και έχουμε όλο και περισσότερα προβλήματα με την αηφορία, με τη βιωσιμότητα, με τους πόρους, ιδιαίτερα με τις ζωοτροφές. Για να μην μιλήσω για τα αντιβιωτικά, για τα δεινά, τα βασανιστήρια των ζώων, για τη διάβρωση του εδάφους. Σωστά τα κατάλαβα Τώρα θέλετε να κάνετε διαφήμιση για να αυξηθεί η κατανάλωση του βοηού κρέατος. Αυτή είναι η λύση στα προβλήματά μας. Αντί να έχουμε ένα μετασχηματισμό σε αυτή την αγορά με μια τοπική γεωργία, μικρή γεωργία, περιφερειακή γεωργία, ακόμα περισσότερο βόη, ακόμα περισσότερες εμπορικές συμφωνίες χρειαζόμαστε. Φτάσαμε στο τέλος του κύκλου των ερωτήσεων. Ε, δεν φαίνεται να ζητά κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο, οπότε να ζητήσω πάλι από τους εκπροσώπους της Επιτροπής να μοιράσετε μεταξύ σας και να ομοδοποιήσετε τις απαντήσεις στις διάφορες ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν. Ε, ευχαριστώ. Η ε, κυρία βέβαια έφυγε. Ρώτησε για τον κανονισμό Omnibus και την ενημέρωσή τους, για την ενίσχυση των γεωργών. Θυμίζω ότι το έχει ξαναπεί στην Επιτροπή Γεωργίας πριν από λίγο καιρό. Και είναι πάρα πολύ ε, σωστό αυτό το επιχείρημα και δεν μπορώ παρά να τονίσω και πάλι τη σημασία που αποδίδουν τα κράτη-μέλη ε, ε, στο να αξιοποιούν καλύτερα ε, τα κράτη-μέλη, οι οργανώσεις παραγωγών και τα λοιπά αυτές τις διατάξεις. Ας πούμε, είδαμε τι έγινε με τους ελαιοπαραγωγούς στην Ισπανία για το ε, άρθρο 2 και πώς το χρησιμοποιούν επιγραμμικά. Είναι πολύ καλή θετική εξέλιξη και ελπίζουμε να έχουμε αντίστοιχες διατάξεις ή αιτήματα. Η αντιπρόεδρο Μαγκίνε αναφέρθηκε στι επιπτώσει των αμέσων ενισχύσεων στην ίδια την Ιρλανδία. Να πω γρήγορα ότι αυτό έχει να κάνει με εσωτερική σύγκληση στην ίδια τη χώρα και καλύτερα να θέσετε την ερώτηση αυτή στις Ιρλανδικές αρχές και όχι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που θα μας ενδιέφερε και εμά να σα απαντήσουμε. Και ε, σε ό,τι αφορά τι εισαγωγέ από την Νότια Αμερική, τι προϊόντα εισάγονται, γιατί θα πρέπει να σταθμίζουμε περισσότερο προς ε, τα ευγενή τα τα φιλέτα ας πούμε και τις μπριζόλες ε, αυτό είναι γεγονός ε, στη Συμφωνία Μερκοσούρ. Θα ήθελα όμως να το ξαναπώ, το είπα και προηγουμένως ε, κάπως ακροθυγός. Το εμπόριο ζωικά προϊόντα και στο βόλιο κρέας θα πρέπει να το βλέπουμε συνολικά ενταγμένο σε ένα πλαίσιο προϊόντων. Για παράδειγμα, όταν μιλώ για οργανώσεις παραγωγών, εμπορε, εμπορικές εξαγωγών, η προτεραιότητά τους στην κινέζικη αγορά είναι ας πούμε, το πουλερικό είναι τα, τα, πόδια των ε, κοτόπουλων που δεν τα, δεν τα αγοράζει κανείς στην Ευρώπη ε, ενώ ε, στην Κίνα ε, πολλούνται αυτά ή τα εντόστια ας πούμε το μοσχαρίσιο το, το βόιο σηκώτη που εδώ δεν το πολυτρώνε αλλά στην Κίνα τρελαίνονται Υπάρχουν και άλλα προϊόντα, πάρα προϊόντα, που δεν σημαίνει ότι είναι κατώτερης ποιότητας, ε, όπου υπάρχει μεγάλο πεδίο δόξης. Ε, σας είπα και προηγουμένως ότι έχουμε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα σε ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς. Αλλιώς αυτά θα τα πετούσαμε τα προϊόντα, ε, θα καταστρέφανε το περιβάλλον. Έχουμε βρει μια πολύ καλή χρήση υψηλής αξίας και πολύ προσοδοφόρα και είμαστε πάρα πολύ ε, ανταγωνιστικοί με πλεονέκτημα και το χρησιμοποιούμε αυτό παγκοσμίω. Αντίστοιχα, όταν μιλώ για ε, χειροτρόφους και τι έγινε με τη Ρωσία, ε, χάσαμε στην ε, εξαγωγή ε, χείριου λίπους που δεν το χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη, στέατος, που ήταν τεράστιο κέρδος αυτό στο παρελθόν που είχαμε πρόσβαση στην Ρωσία. Θα πρέπει να δούμε όλα τα προϊόντα φυσικά. υπάρχουν και τα ευγενή τα μάχια και τα φιλέτα και οι μπριζόλες και τα λοιπά. Ε, φυσικά χώρα, άμα το αναλύσουμε, θα έχουμε νικητές και τιμένους. Στις Ηνωμένε Πολιτείες, ας πούμε, εισάγουν πολύ μεγάλες ποσότητες χαμηλής ποιότητας ε, κρέατος βοήου, γιατί ε, ε, είναι χόρταγη εκεί ως προς τη ζήτηση για τα χάμπουργκερ, ενώ εξάγουν υψηλής ποιότητας φιλέτα και τα λοιπά, τέτοια τεμάχια. στην Ευρώπη, όπως έχουν τα πράγματα σήμερα στο Βόιο, εξάγουμε πολύ περισσότερα από ό,τι εισάγουμε. Μπορεί να χάνουμε σε κάποιες κατηγορίες, αλλά η συνολική εικόνα είναι ότι βγαίνουμε κερδισμένοι από αυτή την υπόθεση. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα που είχε να κάνει με τους Πολωνούς ε, κτηνοτρόφους που ε, έχουν μεγαλύτερες απώλειες από τη Ιρλανδοί και τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα να επεκταθούν. Νομίζω το είπα προηγουμένως. Είπα ότι είναι προς όφελος όλων των ε, γεωργών αυτών και των κτηνοτρόφων, γιατί είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση και η τάση συνολικά σε όλο τον κλάδο. Το Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο προετοιμαζόμαστε για το άτακτο Brexit και οι αγορές ήταν πάρα πολύ ευάλωτες. Και οι βοοτρόφοι περίμεναν ότι μπορεί να έχαναν από τη μια μέρα στην άλλη την πρόσβαση οι Ιρλανδοί και δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην ε, επιρωτική Ευρώπη στην αγορά και κάτι έπρεπε να κάνουμε για να τονώσουμε ε, την εμπιστοσύνη στο Ιρλανδικό Βόλιο. Το κάναμε και αυτό είναι προς όφελος όμως γενικά του κλάδου στην Ευρώπη έγιναν διάφορες ερωτήσεις για το θέμα των ελέγχων γιατί, ε, στους οποίους υποβάλλονται οι εισαγωγές. Ε, κρίμα που δεν υπάρχει συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση σαν να απαντήσει. Ο Επίτροπος Χόγκαν έχει δηλώσει ότι θα πρέπει να είναι δρακόντι η έλεγχη για όλες τις ποσότητες και ισχύει αυτό. Ε, εδώ πολύ συχνά ε, ρίχνουμε το βάρος στη Βραζιλία. Θα ήθελα όμως να τονίσω το εξή και μιλώ μόνο για το Βόιο. Μόνο ορισμένε περιφέρειες στη Βραζιλία ε, έχουν εγκριθεί για εξαγωγές στην Ευρώπη. Κυρίως η τυπική τους πλειονότητα είναι στην κεντρική και νότια Βραζιλία, πολύ μακριά από την Αμαζονία. Και επίσης είναι πολύ λίγες οι εκμεταλλεύσεις που είναι εγκεκριμένες οι εταιρείε. Πάρα πολύ μικρό το κλάσμα λοιπόν της συνολικής ε, ε, παραγωγής βοήου ε, στη Βραζιλία κατευθύνεται προς την Ευρώπη. Το είπα και προηγουμένως, η Ευρώπη παγκοσμίω στην αγορά του βοήου κρέατος δεν είναι πρωταγωνιστής. Οι περισσότεροι παραγωγοί στη Βραζιλία δεν νοιάζονται για την Ευρώπη, αλλά για την Ασία και την Κίνα. Πάντως, οι εισαγωγές προς την Ευρώπη είναι πολύ αυστηρές, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένε και οι περιοχές και οι εταιρείε και ε, κάθε ε, ε, αποστολή, κάθε παρτίδα ελέγχεται, οι φορτωτικές, οι διάφοροι έλεγχοι, γίνονται λογιστικοί έλεγχοι, έλεγχοι ποιότητα στο κρέατος και πολύ σκληρά μέτρα λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Αυτό το λέω σε ένα και μόνο παράδειγμα μια ε, εταιρεία από τη Βραζιλία που είναι του τους ηγέτες παγκοσμίως εξαγωγών, ε, αυτή τη στιγμή έχει βγει από τη λίστα των εγκεκριμένων για την Ευρώπη. Γιατί δεν τηρεί τις προϋποθέσεις. Είναι μάλιστα πολύ αυστηροί. Ε, ζώα χωρίς ορμόνες αυξητικές, χωρίς αντιβιωτικά. Η Ευρώπη είναι πάρα πολύ αυστηρή στους ελέγχους, τους εισαγωγικούς. Και ακόμα και όταν αυτό ε, πυροδοτεί ε, πολύ πικρές και πολύ σκληρές διενέξεις ε, εμπορικές διεθνώς με τους εταίρους μας. Εμείς το οφείλουμε αυτό στους καταναλωτές και στους παραγωγούς μας και δεν τους εκθέτουμε σε αθέμητο ανταγωνισμό για παραγωγή που δεν είναι στις προδιαγραφές μας. Μπορεί να διαφέρουν, αλλά πάνω κάτω αναπερίπτωση, πάντως γενικά εμείς επιβάλλουμε πολύ αυστηρούς κανόνες. Η Αφρικανική Πανόλη του Χείρου και η κατάσταση στην Κίνα σε σχέση με την Αφρικανική Πανόλη του Χείρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα ανώμια πράγματα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Στην Ευρώπη είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στον έλεγχο της Αφρικανικής Πανόλης και τα περισσότερα κρούσματα ε, περιορίζονται ε, σε, ε, στα αγριογούρουνα και σε πολύ λίγους τους χείρους. Στις εμπορικές επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις δεν έχει ξεσπάσει αυτό. Έχουμε στην Ευρώπη ένα πολύ καλό σύστημα ε, βιοασφάλειας και προστασίας της υγείας των ζώων. Δεν σημαίνει ότι δεν επαγρυπνούμε. Φυσικά επαγρυπνούμε και οφείλουμε γιατί σε εμπορικές εκμεταλλεύσεις τα κρούσματα μπορεί να έχουν τεράστια επίπτωση. Και επιμένω Πέντε δις πλεόνασμα έχουμε στις εξαγωγές ε, χοιρινού σε άλλες χώρες του κόσμου. Φανταστείτε, αν σταματήσουν εξαγωγές, θα πρέπει να πουλιέται στην Ευρώπη αυτό. Και θα έχει και τεράστια επίπτωση όχι μόνο στις τιμές, αλλά και για άλλα προϊόντα, το εγώ πρόβιο, το βόιο, το κρέας των πουλερικών κτλ. Εισαγωγές από την Κίνα, ελάχιστες δεν εισάγουμε ούτε χοιρινό από την Κίνα, ούτε βόλιο. Πολύ περιορισμένα εισάγουμε πτηνά, πουλερικά, ε, με πολύ περιορισμένους, ε, περιοριστικούς όρους και κάποιες πρώτες ύλε για παραπροϊόντα, ε, για ζωοτροφές και ζώα συντροφιάς για την Ιρλανδία και τα μέτρα, επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένω. Αυτό δεν το κάναμε για να βοηθήσουμε μόνο του παραγωγού στην Ιρλανδία, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη. Το μέτρο αυτό είναι πάρα πολύ διαφανέ. Είναι νομικό μέσο, είναι δημόσιο, έχει συζητηθεί με τα κράτη-μέλη. Ήταν και μεγάλη αντίδραση σε αυτό το μέτρο και αντίσταση γιατί θα ήθελαν τα κράτη να έχουν τα ίδια μέτρα και δική τους παραγωγή, αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, καταφέραμε να πείσουμε την πλειονότητα των κρατών ότι αυτό θα ήταν προς όφελος όλων των παραγωγών. Ωστόσο θα πρέπει να είμαστε πραγματικά πολύ αυστηροί ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστός ο κανονισμός για την κοινή οργάνωση αγοράς. Ε, υπάρχουν όροι, ε, μια αιρεσιμότητα, οι Ιρλανδικές αρχές είχαν τη δυνατότητα να επιβάλλουν διάφορα μέτρα, παραγωγή, ε, προαγωγή και προώθηση της ποιότητας, περιβαλλοντικά μέτρα. Προφανώς είναι δύσκολη η απόφαση των ελλαδικών αρχών και τους συμπονούμε πραγματικά, αλλά δεν μπορεί να είναι υβριδική η λύση. Εμείς δεν ζητήσαμε μείωση παραγωγής. Εκείνοι επέλεξαν μείωση της εκπομπής νητρικών για ένα χρόνο. Και αυτό αφορά και τους παραγωγούς, αλλά αυτή τη στιγμή περάσει αυτό το διάστημα, μπορούν να επανέλθουν αν θέλουν στην πρώτερη παραγωγή, αν χρειαστεί. Σας βλέπω, Πρόεδρε, ναι, το κατάλαβα το σφυράκι. Ε, για τα θέματα ανταγωνισμού και εμπορίου νομίζω μπορούν να απαντήσουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση τη κύρια Μαγκίνες. Με ρωτήσατε, μπορούμε να επιφύλακτα να πούμε ότι δεν είναι εφαρμόζονται πρακτικές που παραβιάζουν τον ανταγωνισμό στην Ιρλανδία εκ μέρους των μεταποιητών βοηού κρέατος. Όπως θα φαντάζεστε, η απάντηση είναι φυσικά δεν μπορούμε να δηλώσουμε κάτι τέτοιο κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πάντως ότι η εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού προσπαθεί να επιβάλλει Διόλευ καταφρώνει τα πρόστιμα σε περίπτωση που υπάρχει συγκέντρωση καρτέλ. Και μάλιστα ε, το δικαστήριο σχεδόν ε, έκρινε δρακόντια αυτά τα, πρόθυ, αυτά τα πρόστιμα. Οπότε για να κατηγορηθεί κάποιος και να του επιβληθούν τέτοιο σχεδόν εγκληματικά πρόστιμα θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη αυτή η κατηγορία, να υπάρχουν ε, αποδείξεις βάσιμες ε, προκειμένου να διωχθούν οι παραβάτες. Στο παρελθόν επανειλημμένος στο διάλογο που είχαμε με τους Ιρλανδούς παραγωγούς και άλλους ε, συμμετέχοντες στην αγορά είπαμε ότι αν οποιοδήποτε έχει κάποια πληροφορία ή αποδείξεις είτε από καταγγέλλοντα είτε από άλλες ε, πηγές που θα μπορούσε να προκαλέσει έναρξη έρευνα ει βάρο κάποιες εταιρείες και δεν μιλούμε εδώ μόνο για τη γεωργία για την κτηνοτροφία. Είναι υποχρέωση τη πολιτική ανταγωνισμού να δίνεται συνέχεια σε περίπτωση που υπάρχουν κατηγορίε τεκμηριωμένες. Αλλά χωρί αποδείξει, χωρί τεκμήρια, είναι πολύ δύσκολο εμεί να πιθανολογήσουμε αν παραβιάζονται ή όχι αρχέ του ανταγωνισμού. Το ίδιο ισχύει και για τι αρμόδιε αρχέ ανταγωνισμού τη Ιρλανδία, που ήδη έχουν εξετάσει τέτοιες κατηγορίες. Αλλά αν είναι αβάσιμες οι κατηγορίες, δεν τεκμηριώνονται από αποδείξεις, είναι δύσκολο να κινηθεί νομικά μία έρευνα εις βάρος συγκεκριμένης εταιρεία. Και στο παρελθόν, παρελειμμένος οι ενώσεις παραγωγών στην Ιρλανδία είχαν καταγγείλει μια πιθανή συμπεριφορά καρτέλα από μεταπίτες και τελικά έκανε και στον τύπο ανακοινώσει ότι παραπονέθηκα στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και κατήγγειλαν τη σχετική συμπεριφορά. Πάντω, η συγκρότηση καρτέλ είναι μια ιονή ε, εγκληματική δραστηριότητα και υπέχει κάποιο προσωπική ευθύνη και επισύρονται και βαρύτατα πρόστιμα. Οπότε είναι λογικό να γίνεται μια απόπειρα καταστροφή των αποδείξεων. Σβήνονται mail, οποιασδήποτε αποδείξει που μπορεί να τεκμηριώσουν συνάντηση και προσδιορισμό μια κοινή τιμή, τέτοιε αποδείξει εξαφανίζονται. Πολύ εύκολα. Μακάρι να είχαμε αποδείξεις ε, γιατί εμείς πολύ θέλουμε να καταπολεμούμε τέτοιες συμπεριφορές καρτέλ από πλευράς αγοραστών, αλλά για να κάνουμε το καθήκον μας που το κάνουμε πολύ ευχαρίστως, θέλουμε είτε αποδείξεις εκ μέρους, της αρμόδιας, ε, εκ μέρους των καταγγελόντων, ώστε είτε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε οι αρμόδιες Ιρλανδικές Αρχές Ανταγωνισμού να μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία. Οπότε απευθύνω έκκληση προς καταγγέλλοντες, προς επίδοξους καταγγέλλοντες, αν έχουν στοιχεία, ονόματα, έγγραφα που είναι κλειδωμένα σε χρηματοκιβώτια, σας διαβεβαιώ ότι προστατεύουμε τους καταγγέλλοντές μας, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το καθήκον μας, αλλά χρειαζόμαστε αποδείξεις. Σας ευχαριστώ να συμπληρώσω τις ε, ερωτήσεις, τις απαντήσεις. Τι θα γίνει με το βόλιο κρέας της επικείμενες διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία είναι ευαίσθητο προϊόν και σίγουρα θα το διαφοροποιήσουμε σε σχέση με τις άλλες μα εμπορικές συμφωνίες. Προς το παρόν αποκλείεται από τις προσφορές γιατί και εμείς το αντιμετωπίζουμε ως ευαίσθητο προϊόν. Δεν θα υπάρξει άνοιση ή διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με άλλες εμπορικέ συμφωνίες. Σε ό,τι αφορά τη μελέτη ε, βιωσιμότητας και αντικτύπου, παρόλο που η έκβαση των διαπραγματεύσεων του Μερκοσούρ δεν περιλήφθηκε στην μελέτη αντικτύπου, η όλη διαδικασία ξεκίνησε πολύ πριν τη σύναψη της Συμφωνίας Μερκοσούρ. Οπότε είχαμε δύο ε, σενάρια. Το συντηρητικό με περικοπή το 25% των ε, δασμών και το πιο φιλόδοξο σενάριο το 50% περικοπές των δασμών. Και αν δείτε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ε, με τις χώρες Μερκοσούρ, διαπιστώνουμε ότι η δοσμολογική ποσόστοση πλησιάζει προς το συντηρητικό μας σενάριο, προς το 25% περικοπή. Τελικά ε, ήταν 0,7% ε, η μείωση της παραγωγής. Πάντως θα επικαιροποιήσουμε τη μελέτη για το σωρευτικό αποτέλεσμα των εμπορικών συμφωνιών, των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου στη γεωργία και κτηνοτροφία. Και ο υποψήφιο ε, Επίτροπο Γεωργία του υποσχέθηκε στην δημόσια ακρόαση. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις εργασίε. δεν ξέρουμε πότε θα τι ολοκληρώσουμε, πάντως θα πρωτοστατεί σε αυτές η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και εμείς από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου θα προσφέρουμε τη τεχνογνωσία μας για την ολοκλήρωση αυτή τη μελέτη η πραγματική τελικά έκβαση της συμφωνίας Μερκοσούρ θα περιλαμβάνεται στα πορίσματα της νέας μελέτης, της νέας ε, μελέτης αντικτύπου. Επίσης, ε, εξασφάλιση είδων ίδιων προδιαγραφών πρέπει να γίνονται σεβαστές και από τους εταίρους μας. Αυτό το απάντησε ε, ο συνάδελφος Κάνελ, ισχύει για τις τωρινές αλλά και για τις μελλοντικέ μας εμπορικές συμφωνίες. Τα υγειονομικά και φυτογειονομικά μέτρα και τα πρότυπα που απαιτούμε ισχύουν και για τα τοπικά και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Έχουμε τι ίδιε απαιτήσει και εφαρμόζουμε τι ίδιε προδιαγραφέ και στα εισαγόμενα προϊόντα σε ό,τι αφορά τα υγειονομικά, φυτογειονομικά θέματα. Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Υπάρχει ε, στην Συμφωνία Μερκοσούρα ένα κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα του εμπορίου που καλύπτει τη δέσμευση των χωρών κυρίως των χωρών Μερκοσούρ και φυσικά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη Συμφωνία των Παρισίων που σημαίνει από πλευράς Μερκοσούρ και κυρίως Βραζιλίας ε, μηδενική παράνομη υλοτομία η αποψήλωση και η υποχρέωση αναδάσωσης 12 εκατομμυρίων εκταρίων. Αυτή την δέσμευση την έχει ήδη αναλάβει η Βραζιλία. Μάλιστα ακόμη και αν ο πρόεδρος της Βραζιλίας αποσυρθεί από τη Συμφωνία των Παρισίων, αυτό θα σημαίνει όχι μόνο παράβαση της Συμφωνίας των Παρισίων, αλλά αυτόματη ε, καταστρατήγηση και της ε, Συμφωνίας Μερκοσούρ, με τις συνέπειες που θα έχει κάτι τέτοιο. Αναφέρθηκε λοιπόν το περιβάλλον. Το κεφάλαιο βιωσιμότητα και οι περιβαλλοντικέ ε, υποσχέσει υπόκειται στη διαδικασία διακανονισμού των εμπορικών διαφορών και υπάρχει κάτι ειδικό για το περιβάλλον που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να παραχθούν αποδείξεις ότι υπάρχει βλάβη ε, στο περιβάλλον, ζημία στο περιβάλλον, που κάτι που απαιτείται για άλλου είδους ε, διακανονισμό στις εμπορικές ε, διαφωνίες. Επίσης, τα υγειονομικά, φυτογειονομικά μέτρα ισχύουν και για τα περιβαλλοντικά θέματα. Δηλαδή, αν χρειάζονται μέτρα θα ληφθούν εφόσον δίνονται απαραίτητε πληροφορίε και επικαιροποιημένε. Αυτό είναι γνωστό για τα φυτογεωνομικά μέτρα και το επεκτείνουμε και στα περιβαλλοντικά κεφάλαια της συμφωνίας. Και τέλος, ως προς την ερώτηση με τι βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιορίζει και καθορίζει τις δασμολογικές ποσοστώσεις, αυτό γίνεται περιπτωσιολογικά και ανάλογα με τον εταίρο μας. Πάντως, δεδομένη της ε, σύναυσης της ε, συμφωνίες που συζητούμε αλλά και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, ένας από τους στόχους της σωρευτικής μελέτης ήταν να έχουμε μια ιδέα του αντικτύπου. Και λαμβάνουμε, λαμβάνουμε υπόψη τον αντίκτυπο με το συγκεκριμένο εταίρο και όλα αυτά τα στοιχεία τα συμπεριλαμβάνουμε στην ανάλυση των προσδιορισμό και το σχεδιασμό των πιθανών δασμολογικών ποσοστώσεων για τη συγκεκριμένη, επαναλαμβάνω, εμπορική συμφωνία για την οποία έγινε και μελέτη αντικτύπου. Ευχαριστώ. Yeah, vielen, vielen Ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την τόσο ευρεία παρουσίαση. Ε, τα στοιχεία υπάρχουν και για τα μέλη ούτως ή άλλως. Ε, ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήρα μέρος στην όλη συζήτηση γιατί όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την ε, παραγωγή ε, βοηού στην Ευρώπη και για την κτηνοτροφία. Ο κύριος Γιουρκέλ. Κύριε Πρόεδρε, δεν απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα γίνει μια εξίσωση των άμεσων ενισχύσεων για να αντιμετωπιστεί η κρίση ή τουλάχιστον θα δοθεί μια αντιστάθμιση, αποζημίωση στους γεωργούς και παραγωγούς και κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από αυτή την ε, ανισότητα των άμεσων ενισχύσεων. Δεν απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. To come again, but... Θέλετε να απαντήσετε και πάλι, να πάρετε το λόγο, αλλά πάρα πολύ γρήγορα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το μέτρο που αναφέρατε ήταν έκτακτο μόνο για την Ιρλανδία και τους Ιρλανδούς παραγωγούς όμως τα, τα παράλληλα αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα για τους άλλους Ευρωπαίους παραγωγούς, τη συντηρητική τους πλειοψηφία στα κράτη-μέλη, Υπήρξε αλληλεγγύη και υποστηρίχθηκε αρχικά. Δεν υπήρξε επίση πρόταση να παραταθεί και να σχέσει περαιτέρω. Εάν υπάρξει ανάγκη στι αγορέ, θα χρειαστεί να παρέμβουμε και να στηρίξουμε την αγορά στην Πολωνία, τη Δημοκρατία τη Τσεχία, στη Σουηδία, ξέρω εγώ, αναλόγω πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά ο συγκεκριμένο κανονισμός είχε σκοπό να αντιμετωπίσει αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση εκτάκτος. Ωραία. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε διάλογο. Μπορείτε και δημερός να τα δείτε λεπτομερέστερα. Ολοκληρώνουμε την εξέταση του σημείου αυτού λοιπόν, του 9ου και περνάμε στο 10 λιγότερο συναισθηματικά φορτισμένο από ότι το προηγούμενο, θέσπιση προγράμματο για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων και τι ευρωπαϊκέ στατιστικέ. Η υπεύθυνη επιτροπή, η καθήλυνα αρμόδια είναι η ΙΜΚΟ εμείς συμμετέχουμε ως Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη της Υπέθρου. Υπάρχουν κάποια προγράμματα όπως τη διατροφικής αλυσίδας που ε, έχουν κάποια σημασία για μας. Την αρμοδιότητα λοιπόν για αυτά τα θέματα έχουμε εμείς. Ε, η είναι η κυρία Σμιτ Μπάουερ και μπορεί να μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου τριμερούς διαλόγου το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πρόεδρε συνάδελφοι να σας ενημερώσω για τον πρώτο τριμερή διάλογο Καταρχάς, να, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους ως τώρα και τη δουλειά τους στο θέμα αυτό και έχουμε τα σχετικά έγγραφα μπροστά μας. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έλαβε χώρα στο τελευταίο Στρασβούργο. Συζητήσαμε πρώτα απ' όλα για τις πολιτικές προτεραιότητες που θα πρέπει να δώσουμε στις δημοτεύσεις, μετά κάποια τεχνικά σημεία σε τεχνικό επίπεδο και επίσης είδαμε και το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Όπως είπατε, καθήλυνα αρμόδια είναι Επιτροπή Περιβάλλοντος και προστασία του Αναλωτή, όμως εδώ έχουμε κάποιες αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΙΜΚΟ και μετά έχουμε κάποια μέτρα που αφορούν τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και τομές που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών ή την ε, υγεία των ε, φυτικών προϊόντων. Εδώ λοιπόν μας απασχολούν κάποια θέματα πρόληψης, μέτρα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων κρίσης και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Σημαντικό είναι το πρόγραμμα αυτό να αναπτυχθεί περαιτέρω στα πλαίσια της αηφορίας με προϊόντα αηφορίας και τη χρήση ε, των τροφίμων με προσθές τιμές. Επίσης καινοτομία είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Και τι μπορεί να γίνει με τα μέτρα στήριξης της οικονομίας για τον τομέα παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών. Επίσης, για την προστασία των φυτικών προϊόντων και των φυτών πρέπει να υπάρξει κατάλληλη χρηματοδότηση. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα τρίτο του συνολικού προγράμματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα της τροφικής αλυσίδας και των τροφίμων θα πρέπει να προβλέψει ένα αποθεματικό της κρίσης, ένα λεγόμενο emergency reserve, ε, για να αντιμετωπίσουμε μελλοντικέ κρίσει. Αυτό το έχει προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο άρθρο 12 για όσου ενδιαφέρονται στο πρόταση για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο και σε περιπτώσεις κρίσεων, ένα τέτοιο αποθεματικό, ένα τέτοιο ταμείο θα μας επιτρέψει να αναλάβουμε μέτρα υγειονομικά και φυτο ώστε να αντιμετωπίσουμε πιθανά προβλήματα. Αυτό για την υγεία και των ανθρώπων αλλά και των φυτών. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μάλλον, συγγνώμη, η Επιτροπή Γεωργίας θέλει να δει και τον περιορισμό των τη πράξεων και των εκτελεστικών. Είναι σημαντικό ε, για, τον, για την κατεύθυνση των παρών ή διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια, την συνάδελφο Σμιτ Μπάουερ. Υπάρχουν ερωτήσεις προς την εισηγήτρια. Όχι. Οπότε λαμβάνουμε γνώση τη πρόοδου των διαπραγματεύσεων και σα ευχόμαστε καλή τύχη για τη συνέχεια των τριμερών διαλόγων. Και τώρα πάμε απευθεία στο σημείο 11. Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ιστορικό. Ξέρετε συνάδελφοι ότι 5 Νοεμβρίου σήμερα 2019 είναι σαφές ότι δεν βρεθήκαμε στη θέση να ολοκληρώσουμε, να περατώσουμε τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, ιδίως με το στρατηγικό σχεδιασμό των κρατών μελών, ώστε 1η Ιανουαρίου 2021 να είναι όλα ε, έτοιμα να ξεκινήσουν. Ε, χρειάζεται και χρόνο ούτως ή άλλως εδώ για να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, περιμένουμε εδώ και καιρό να κάνετε σχετικές προτάσεις. Εδώ 31 Οκτωβρίου, πριν από ελάχιστες μέρες, είχαμε τις πρώτες δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία περισσότερα τεχνικού χαρακτήρα, η πρώτη, και μια δεύτερη πρόταση πολιτικός περισσότερο ενδιαφέρουσα για μας, με περισσότερες πολιτικές πτυχές και τα είδαμε και σήμερα στην σχετική συνεδρία των συντονιστών. Αναθέσαμε μάλιστα έκθεση και ανέλαβαν οι αρμόδιοι. Αυτά ως προς την ε, τωρινή κατάσταση των πραγμάτων. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε αναλόγως να μας παρουσιάσει τις προτάσεις της, ο λόγος στον κύριο Νίγια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και μέλη του Κοινοβουλίου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι προτάσεις για τη μετάβαση αναμένονται διακαώς και από τους δύο συνομοθέτες, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που σήμερα θα είμαι σε θέση να σας τα παρουσιάσω. Εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους την περασμένη Πέμπτη. Όπως θα δείτε ήδη από την πρώτη πρώτη διαφάνεια, σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την συνέχεια ε, προστασίας των γεωργών και κτηνοτρόφων από την ΚΑΠ και μετά το 2021. Θα επανέλθω σε λίγα λεπτά για να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για την ε, συλλογιστική που οδήγησε στην πρότασή μας. Πρώτα όμως να σας πω λίγο το ιστορικό της όλης πρότασης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θυμίσουμε ότι μια ταχεία συμφωνία για τις προτάσεις μεταρρύθμισης ε, της ΚΑΠ παραμένει προτεραιότητα για μας. Αυτό περιμένουν και οι δικαιούχοι της ΚΑΠ. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, πολύ εύστοχα, ότι όταν δούμε το σημερινό προγραμματισμό δεν φαίνεται να είναι πια ε, εφικτό να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία για τα στρατηγικά προγράμματα της ΚΑΠ ε, και ώστε να εφαρμοστούν αυτά από τα κράτη-μέλη 1 Ιανουαρίου του 2021. Αυτό έχει προτείνει αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απίθανο πλέον. Έτσι νομίζαμε το 2018 στις προτάσεις μας βασιστήκαμε στην υπόθεση ότι τα κράτη-μέλη θα χρειαστούν τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις εσωτερικές διαδικασίες έγκρισης των σχεδίων τους και να τα εγκρίνει εγκαίρως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να αντιστρέψουμε λοιπόν τους χρονικούς υπολογισμούς, θα πούμε ότι οι προτάσεις μας δεν δίνουν το επιθυμητό χρονικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό φαίνεται ότι θα είναι έτος μετάβασης το 2021 και θα γίνει αυτό για ένα χρόνο γιατί και πάλι ελπίζουμε ότι οι συνομοθέτες θα προλάβουν ως τότε. Θα καταφέρουν να συμφωνήσουν κάπου το ερχόμενο καλοκαίρι. Έχοντας το λοιπόν αυτό κατά νου, ελπίζουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα ξεκινήσουμε τουλάχιστον με τα στρατηγικά σχέδια εξού και το έτος μετάβασης. Ε, Ενάμιση χρόνο πάλι. Από την επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι επιτάπητο έχουμε δύο νομοθετικέ προτάσει. Ο λόγος που τα χωρίσαμε σε δύο είναι γιατί έχουμε διαφορετικές χρονικές, ε, χρονικούς ορίζοντες για τις δύο προτάσει. Η πρώτη είναι ο κανονισμό ευελιξίας, όπω ονομάστηκε, ελαστικότητας, άκρο τεχνικό, με τρεις ε, βασικές αλλαγές. Πρώτον, να κοιτάξουμε να διασφαλίσουμε την συνέχεια μεταξύ της στήριξη της ΚΑΠ στα ημερολικά έτη 2020 και το δημοσιονομικό το 2021. Το 2020 ήδη υπήρχε πρόταση που είχε ζητηθεί από τους συνομοθέτες να εγκρίνουν στην τακτική νομοθετική διαδικασία μέχρι τα τέλη της περσινής χρονιάς ο λεγόμενος κανονισμός 2020 και εκεί χρησιμοποίησαμε τη διαδικασία fast track για να προλάβουμε γρήγορα. Οι κανόνες εκεί πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να λάβουν υπόψη κάποιε δυσκολίε που ανακαλύψαμε, κυρίω στην ευελιξία μεταξύ των ε, πυλώνων. Και μετά, το δεύτερο που είναι πιο σημαντικό, εκεί έχει ένα σωρό κανόνε και φανταζόμαστε ότι υπάρχουν συζητήσει συζητήσεις και υποβολέ τροπολογιών από του δύο συνομοθέτε. Εκεί σκεφτήκαμε ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος στη διαδικασία συνομοθεσία και ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί ω το καλοκαίρι του 2020 από του δύο συνομοθέτες. Για το πρώτο όμω, Είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θέλουμε να εγκριθεί. Αυτό ελπίζουμε. Για μια σειρά από λόγους ε, μπορεί να είναι εφικτό, άντε μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους. Ο πρώτος λοιπόν ε, κανονισμός που είναι και πολύ σύντομος, ο κανονισμός της ευελιξίας, της διαλεκτικότητας. Ε, επικαιροποίηση των όρων αναφοράς για την δημοσιονομική πειθαρχία και μετά και ένα θεματάκι για τη μεταφορά μεταξύ πυλώνων. τον παλιό λεγόμενο κανονισμό του 2020 έχουμε μια σχετική διάταξη που όμω δεν λειτουργήσε αποτελεσματικά και δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρί το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό ήταν ένα λόγο. Όπου τα κράτη-μέλη που θα θελήσουν να μεταφέρουν κονδύλια στι απευθεία πληρωμέ από την ανάπτυξη υπαίθρου για το αμερολογικά του 2020 θα χρειαστούν αυτόν τον ειδικό κανόνα. Αυτό δεν θα βασιστεί σε ποσοστά πλέον, αλλά σε μέγιστα απόλυτα ποσά, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορεί να ε, εφαρμοστεί. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι ως το τέλος της χρονιάς και μέχρι τις αρχές της επόμενης, όταν υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχει εγκριθεί ο κανονισμός αυτός, δεν θα έχουμε ακόμη την συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το σύνολο του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου για ολόκληρη την περίοδο. Και μετά υπάρχει και μια άλλη πολυτεχνική λεπτομερία, δηλαδή η ρήτρα αναθεώρηση από τα κράτη-μέλη των ποσών για την ΚΑΠ για το 2020. Όπω είπα, είναι άκρο τεχνικό όλο αυτό και ελπίζουμε ότι οι δύο συνομοθέτε θα το συμφωνήσουν και θα τα βρουν με μια διαδικασία fast track τρόπον ά, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να το εφαρμόσουν ε, ήδη στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Και μετά έχουμε μια ένα μεγαλύτερο, ευρύτερο κανονισμό μετάβαση και έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά και πάλι είναι φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα, το παραδέχομαι. Εδώ τι περιλαμβάνονται τα θέματα που βλέπετε στις διαφάνειες, αλλά κυρίως ε, βασιστήκαμε στη, συλλογική, στη λογική ότι θέλουμε τη συνέχεια της ΚΑΠ ε, και τη συνέχεια μεταξύ των δύο πυλώνων, ανάπτυξη τη υπαίθρα, πληρωμές συνδεδεμένες πληρωμές, ε, τομεακές και μέχρι το 2021, εφόσον ε, βασιστούμε στους κανόνες που είχαν εγκριθεί και από το Συμβούλιο και εσά το 2013. Ένα σημείο θέλω να τονίσω εδώ, ότι θέλουμε να συμπεριλάβουμε όλα τα προγράμματα δαπανών και όπως ξέρετε όλοι οι κανονισμοί επιτρέπουν να πάρουμε κονδύλια στα παρατήματα το λέει αυτό, αλλά και στο σώμα του κειμένο μέχρι το 2020, αλλά και το 2021. Γιατί το 2021 είναι η πρώτη χρονιά. Η πρώτη χρονιά του πολιτός δημοσιονομικού πλαισίου, που για την ώρα δεν έχουμε καθόλου αριθμού. Οπότε ο κανονισμό αυτό ε, δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη, ακόμη και αν επισήμως εγκριθεί, διότι δεν θα έχουν τα ποσά για να τα εκταμιεύσουν και να τα στείλουν στου δικαιούχου. Οπότε υπάρχει αυτή η λακούνα, αυτό το κενό που θα πρέπει να το καλύψουμε κάπως και γι' αυτό οι κανονισμοί μετάβασης προβλέπουν σε διαφορετικά τμήματα των παρατημάτων να πάρουμε κάποια κονδύλια για το 2021. Θα αναρωτηθείτε βεβαίω, δεν έχουμε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τι βάση την κάνει την πρόταση αυτή. Οι αριθμοί που θα δείτε στην πρότασή μα είναι υποθετικοί. Βασιζόμαστε στην πρόταση για το, δημοσιονομικό, για το πούδο που από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ε, έπρεπε κάπω να ετοιμάσουμε την πρότασή μα για να ξεκινήσει η διαδικασία τη συνομοθεσία. Και Βασιστήκαμε στου αριθμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Πουδουπού. Εδώ λοιπόν βασιστήκαμε στην υπόθεση εργασία ότι μέχρι του χρόνου που ο κανονισμό αυτό θα πρέπει να έχει εγκριθεί από του δύο συνομοθέτε, θα έχουμε πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και τότε βεβαίω θα μπορέσουν οι δύο συνομοθέτε λογικώ να αντικαταστήσουν του αριθμού που έχουμε βάλει εμεί στην πρότασή μα με του σωστού. Αυτού που τελικώ θα συμφωνήσουν. Άλλοι θα έλεγαν ότι τεχνικώ όλα αυτά θα έπρεπε να μπουν σε αγγείλε, γιατί είναι μια υπόθεση εργασία ούτω ή άλλω, αλλά τέλο πάντων έτσι προσεγγίσαμε την όλη πρόταση. Και μετά υπάρχουν κάποιε προσαρμογέ για να βεβαιωθούμε ότι οι κανονισμοί μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν σωστά και το 2021. Ταυτόχρονα, έχουμε, και αυτό ισχύει κυρίω για τα τομεακά προγράμματα, την εξή δυσκολία κάποια από τα τομεακά προγράμματα για τον Ίνο, τα παρακυπευτικά, τη Γεωργία. Ε, αυτά προτείναμε να μεταφερθούν από τον τωρινό κανονισμό για την ΚΑΠ στα στρατηγικά ε, προγράμματα. Όμως κάποια από αυτά έχουν διαφορετικό χρονικό ορίζοντα. Κάποια ξεκινάνε πριν από το 2022, κάποια ξεπερνάνε το 2022. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε βάσει κάποιων κανόνων να δούμε πόσο τα παλιά προγράμματα μπορούν να παραταθούν ε, στην τωρινή τους μορφή και ε, πότε μπορούν να ενταχθούν στα στρατηγικά προγράμματα της ΚΑΠ. Για να το συντομεύω. Αυτό που προτείνουμε είναι να κλείσουν τα προγράμματα αυτά, αυτά που ολοκληρώνουν πριν την 1η Ιανουαρίου 2022 και να παραταθούν για μια πολύ σύντομη χρονική περίοδο για να ενσωματωθούν πλήρω από την 1η Ιανουαρίου 2022 στα στατηγικά προγράμματα τη ΚΑΠ. Ενώ για τα άλλα προγράμματα που έχουν μεγαλύτερο κύκλο ζωή, αυτά μπορούν να συνεχίσουν εφόσον ολοκληρώνονται το 2022 ή 2023. 23. Ε, Εκπνέουν και μετά περνάμε απευθεία στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Και μετά κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την μεταφορά προηγούμενων ποσών για τις δαπάνες από τα στρατηγικά προγράμματα. Τώρα, Στη διαφάνεια αυτή έχετε τις λεπτομέρειες της πρότασής μας. Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες τώρα, δεν είναι καλή ιδέα. Τα βλέπουμε σε άλλη φάση. Απλώς να δούμε δύο-τρία βασικά στοιχεία. Αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια είναι ότι θα επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να παρατείνουν τα προγράμματα ανάπτυξη τη υπαίθρου στην τωρινή του μορφή για, για το μεταβατικό έτο 2021. Ταυτόχρονα όμω θεωρούμε ότι η δυνατότητα αυτή πρέπει να προσφερθεί μόνο στα κράτη-μέλη που πραγματικά μπορούν να ξεμείνουν από κονδύλια. Δηλαδή παλιό χρήμα που στερεύει και εφόσον δεν μπορούν να τηρήσουν τι δεσμεύσει του το 2021 προ του δικαιούχου γιατί δεν έχουν χρήμα, εκεί θα υποστηριχθούν. Κάποια άλλη κράτη-μέλη όμω έχουν ένα μεγάλο πλεόνασμα που θα μπορούσαν να το ξοδέψουν, να το δαπανίσουν από την προηγούμενη περίοδο και για αυτού προτείνουμε να εφαρμόσουν να εκταμιεύσουν δηλαδή το παλιό χρήμα, αυτά τα προηγούμενα κονδύλια, βάσει των παλιών κανόνων. Στην περίπτωση παράταση ε, προγραμμάτων για την ανάπτυξη τη πέθου του 2021, θα προσφερθεί δυνατότητα αυτή μόνο σε όσου έχουν ήδη εξοδέψει όλα τα ποσά από την τωρινή περίοδο και το 2021 μπορεί να ξεμείνουν και δεν θα μπορούν να τηρήσουν νέε δεσμεύσει. Εδώ λοιπόν υπάρχει ιεράρχηση. Όπου υπάρχει παλιό χρήμα, τα κάτι μέλη πρέπει πρώτα να το ξοδέψουν και για όσους το έχουν ήδη ξοδέψει να παρατείνουν τα προγράμματά τους. Βάσει των παλιών προγραμμάτων να εξοδέψουν νέο χρήμα το 2021. Όπως βλέπετε υπάρχουν κάποιες τεχνικές προσαρμογές εδώ, απαραίτητες, για να βεβαιωθούμε ότι εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες για τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου το 2021 για τις απευθείς πληρωμές. Υπάρχει κάτι που το ονομάσαμε ρήτρα αμνηστίας. Δηλαδή, για το, από την 1η Ιανουαρίου 2020 τα δικαιώματα που θεμελιώνουν οι γεωργικοί κοινοτρόφοι πρέπει να θεωρηθούν νόμιμα και τακτικά ε, εφόσον υπήρξαν στο παρελθόν αβεβαιότητες τώρα μπορούν να έχουν αυτά τα δικαιώματα και να τα ασκήσουν και τεχνικές πάλι διθετήσεις για να υπάρξει για το 2021 το έτος ε, που θα προκύψουν οι αξιώσεις του χρόνου ε, να υπάρξει μια ευελιξία μεταξύ των πυλώνων σημαντική κυρίως για τα νέα Το σύστημα SAPS, ε, σύστημα ενιαίος πληρωμής ενιαίας έκτασης πληρωμής θα ισχύσει και για το 2021 με ενιαίους λογαριασμούς. Όπως το είχαμε ε, προβλέψει και στις προτάσεις ε, τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ, ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη που θέλουν να εφαρμόσουν το σύστημα ΣΑΠΣ. Και μετά κάτι που το ανέφερα στην κατηγορία των τομεακών θεμάτων. Κάποια προγράμματα που λίγο νωρίτερα θα παραταθούν για λίγο, κάποια που ε, λίγο, λίγο μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 θα μπορούν να, να, διαρκέσουν λίγο παραπάνω και μετά να ενταχθούν στα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. Μετά κάποιες τεχνικές προσαρμογές στον οριζόντιο κανονισμό, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να αναπτυχθεί στην παρουσίασή μου σήμερα το απόγευμα. Με αυτά και με αυτά να κλείσω και να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσά, κύριε Νίγερ. Θα πρότεινα τώρα να ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές σε ένα πρώτο γύρο και στη συνέχεια τους υπόλοιπους συναδέλφους που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Ο συναδέλφος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός, όπως είπε και ο κύριος Νίμαϊερ, ε, Νίγερ, συγγνώμη, ε, έχουν έρθει ε, αργά αυτά τα κείμενα τα περιμέναμε νωρίτερα. Σήμερα στη συνεδρίαση ε, των ε, συντονιστών αποφασίσαμε να δουλέψουμε γρήγορα και προτείνουμε ε, τον πρώτο κανονισμό να τον διεκπαιρεώσουμε πολύ γρήγορα και για το δεύτερο να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος πολιτικά. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Είναι γεγονός, η δεύτερη η πρόταση κανονισμού είναι απλώς μεταβατική, αλλά έχει ε, πολιτική σημασία γιατί οδηγεί άμεσα στα στρατηγικά σχέδια, ε, τα οποία εδώ στο Κοινοβούλιο όμως δεν έχουν ε, αποφασιστεί ποτέ. Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα ούτε εδώ στο Κοινοβούλιο ούτε με τα κράτη-μέλη. Και αυτό δεν το θεωρώ και τελείως έτσι χωρίς προβλήματα. Έχω μια ειδική ερώτηση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Πρώτον, σωστά το κατάλαβα υποθέτεται ή θεωρείται ότι για τις πληρωμές για το 2021 ε, έχουμε ως αφετηρία την πρόταση του Επιτρόπου Ούτιγκερ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το δεύτερο πυλώνα όμως αυτό έχει βαρύνουσα σημασία γιατί προβλέπει μεγάλες περικοπές εκεί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όπου η χρηματοδότηση του δευτέρου πυλώνα έχει εξαντληθεί. Και τώρα το 2021 έχουν ε, πολύ λιγότερα ποσά για να τα βγάλουν πέρα και να συνεχίσουν τα εφιστάμενα προγράμματα. Ε, πράγμα που ε, ενδεχομένω να δημιουργούσε δυσκολίε. Σωστά είπατε κύριε Νίγιαρ ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν αν θα έχουν χρήματα για να συνεχίσουν τα προγράμματα στο δεύτερο πυλώνα, αν χρειάζονται φρέσκο χρήμα. Αυτό ποιος θα το αποφασίσει, τα κράτη-μέλη, ε, σε επίπεδο κρατικό ή και σε επίπεδο περιφερειών, γιατί έχουμε πολλά κράτη-μέλη ε, που ε, είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση, ιδιαίτερα για την Ήπεθρο. Και υπάρχουν περιφέρειες που δεν έχουν χρήματα για τα σχέδιά τους, ενώ κάποιες άλλες δεν τα έχουν ακόμα ακουμπήσει. Ευχαριστώ. Ε, ο συνάδελφος ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα μας φέρνει τις νομοθετικές προτάσεις της. Να το θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους. Ε, το ζητάμε από τον Ιούνιο. Έχουν περάσει έξι μήνες. Αυτές τις νομοθετικές πράξεις τις παρουσιάζει τώρα Νοέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει λοιπόν να βιαστούμε και να τις εγκρίνουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα, αλλά ως προς το χρονοδιάγραμμα του Κοινοβουλίου θα έλεγα ότι το βρίσκω από την πλευρά της Επιτροπής τουλάχιστον λίγο περίεργο. Ε, όπως είπε και ο κύριος Ντόρφμαν λοιπόν και σε ό,τι αφορά τα θέματα της μετάβασης πρέπει να κατανοήσουμε πώς ακριβώς θα συμπληρωθεί η διαδικασία τρεις νομοθετικές πράξεις που συζητάμε ε, για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Στη φάση αυτή ε, πρόκειται να λάβουμε αποφάσεις για συγκεκριμένα άρθρα με παρεμβάσεις μας. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Δεν θα αρκέσει λοιπόν ένας χρόνος. Το λέω ξεκάθαρα. Θα χρειαστούμε περισσότερο καιρό. Ε, και αντιστρόφω για ο κανονισμό τη ευελιξία μεταξύ των πυλώνων, και μπορούμε να πάμε και με στραπία ταχύτητα. Με μια έγκριση εφόσον πρόκειται για κανονισμό. Αστραπή, εφόσον πρόκειται για κανονισμό ακροστεχνικό. Αλλά η όλη συζήτηση για την ΚΑΠ δεν μπορεί να βιαστεί. Θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά και, σκέφτον, και καλό όλου του συναδέλφου να το πράξουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Νάβατσεκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβολή των προτάσεών της γιατί είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μεταβατικές διατάξεις και είναι η μόνη λύση αυτή η πρόταση που εξασφαλίζει κάποια προβλεψιμότητα για τους γεωργούς μας μέχρι ότου συμφωνηθεί η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Δεν θα επαναλάβω τα σχόλια των συναδέλφων γιατί Πιστεύω και εγώ ότι δεν είναι τεχνικό μόνο το θέμα, ούτε αυτόματο. Υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα. Και η μεταφορά διατάξεων από μία περίοδο στην άλλη θα γύρει πολλά τεχνικά και άλλα ζητήματα που θα κληθούμε να τα συζητήσουμε. Λυπάμαι όμως για την πρόταση για, τις... για την κατανομή των κονδυλίων. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προεξοφλεί τη Συμφωνία Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έτσι φαίνεται από τι προτάσει που κάνει. Η πρόταση όμω για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχει εγκριθεί ακόμη για πολλά κονδύλια και ιδιαίτερα για αυτό τη αγροτική ανάπτυξη, γιατί προϋποθέτει πολλές περικοπές. Οπότε δεν θα πρέπει να προδικάζουμε να προεξοφλούμε μια συμφωνία που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί χρειάζονται πολύ περισσότερες συζητήσεις. Ευχαριστώ κύριε Σχόισλινγκ. Ε, ουσιαστικά ήταν τελείως λογικό να χρειαζόμαστε μια μεταβατική περίοδο. Από πέρσι το συζητάμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι πρόσφατα ισχυριζόταν ότι δεν χρειαζόταν και ότι είναι εντάξει η ΚΑΠ και γρήγορα θα τα βγάλουμε πέρα. Αυτό ήταν τελείως ε, ανεδαφικό. Και τώρα ε, με, το να βασίζεστε στην πρόταση Oettinger με ανησυχεί γιατί σίγουρα ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι το τελικό προϊόν των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Σιώτιγκερ ο ίδιος έκανε μια πρόταση που δεν μπορεί να γίνει δεκτή εδώ. Το είπε ο κύριος Ντόρφμαν για τις περικοπές στο δεύτερο πυλώνα. Ε, οπότε όλα αυτά κάπως με θορυβούν και με ενοχλούν. Και είπατε όσοι έχουν χρήματα να, τα, να συνεχίσουν να τα δαπανούν. Αυτοί που τα έχουν εξαντλήσει, πού θα βρούνε τώρα, ε, θα έχει νέο χρήμα. Και το είπε και ο κύριος Δεκάστρο στη Γερμανία. Έχουμε 16 ομόσπονδα κρατήδια που έχουν ξεχωριστά προγράμματα για το δεύτερο πυλώνα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, θα πρέπει να τα λάβουμε όλα υπόψη. Και μετά... Τώρα ε, κάνει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εκπονεί σε μια μεταβατική περίοδο. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Προφανώς και δεν θα διαρκέσει ένα χρόνο, αλλά δεν μπορούμε και αρον άρων τώρα μέσα σε λίγες εβδομάδες να το περάσουμε. Ε, δεν ξέρω αν ήταν πολιτική επιδίωξη ε, και πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πιέσει πριν τις εκλογές. Ε, αλλιώς αποκοιμήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω. Δεν φταίμε εμείς τώρα αρχίστε να μας τριμώχνετε. Θα κάνουμε τη δουλειά μας με την ησυχία μας και με το χρόνο που χρειάζεται. Ευχαριστώ, κύριος Ντάβιτ. Και εγώ πιστεύω ότι οι συνάδελφοι έχουν δίκιο. Και με κάλυψαν στα ουσιώδη. Οπότε δεν έχω άλλα σχόλια. Ο κύριος Κουσμιούκ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, βέβαια, οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο κανονισμό, που είναι τεχνικός, εντάξει, μάλλον θα είμαστε σε, σε θέση να τον ε, εγκρίνουμε πολύ σύντομα. Μάλιστα, οι συντονιστές αποφάσισαν να το αναλάβει ο Πρόεδρος, οπότε θα τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση. Αλλά έχουμε και δεύτερο κανονισμό και μετά την παρουσίαση καταλάβαμε πόσο περίπλοκος είναι και πόσες ε, συζητήσεις θα χρειαστούν. Κάτι που θα είναι και πιο χρονοβόρο. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι στα μέσα του χρόνου θα έχουμε το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα κράτη-μέλη θα έχουν πια νούμερα και συγκεκριμένα κονδύλια που θα προκύπτουν από αυτή τη συμφωνία για το πιδελταπή. Αλλά δεν είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και οι δημοσιονομικές προοπτικέ για το 2021 και 2027 πολύ πιθανόν να περιμένουν το τέλος του 2021 για να εγκριθούν. Και τότε τι γίνεται. Νομίζω ότι η υπεραισιοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι, αν μη τι άλλο, αδικαιολόγητη. Ευχαριστώ, κύριος Φλάναγκαν. Υπόθηκαν ήδη. Τέλεια. Γλιτώνουμε και χρόνο. Περνάμε στου υπόλοιπου ομιλητέ ο κύριο Κρίστενσεν. Ευχαριστώ, θα τα πω δανέζικα. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευχαριστούμε που μας υποβάλλατε τις προτάσεις αυτές. Είναι σημαντικό για τους Ευρωπαίους γεωργούς και εκτινοτρόφους να γνωρίζουν ότι προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος και να μπορούν να στηριχθούν σε αυτή την προοπτική. Αλλά γιατί προτείνεται ένα μόνο χρόνο. Δεν νομίζω να είναι εφικτό. Δεν νομίζω να γίνονται όλα αυτά μέσα σε ένα χρόνο. Ε, θα ήταν καλύτερα να επιδιώξουμε ποιότητα παρά ταχύτητα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αμάρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, υπόθηκαν αρκετά, αλλά ούτε εγώ συμμερίζομαι την αισιοδοξία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπω οι συνάδελφοι. Δεν θα φτάσει ένα χρόνο. Παρά όμω την ε, καλή δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να πω εδώ και το εξή. Και θέλω να το τονίσω. Δεν θα ήταν και ένδειξη σεβασμού προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήδη έχει τοποθετηθεί για τα θέματα αυτά να δεχτεί μια μεταβατική περίοδο με αξίε για την πρόταση μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού να το δεχτούμε αυτό. Και ρωτώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλά γιατί η χώρα μου δεν το συζητάω καν. Ε, αλλά πώ προδικάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα εφαρμοστούν αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μπορεί να τα εφαρμόσει, αλλά το Κοινοβούλιο όχι. Το βρίσκω λοιπόν τεράστια αδικία να υπάρξει αυτή η υποχρεωτική μεταβατική περίοδος στα ένα ή τα δύο χρόνια. και με απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς τις προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν ήταν δίκαιο να χρησιμοποιηθούν λοιπόν οι αξίες μιας μεταρρύθμισης στα πλαίσια ενός πουδοπού, ενός πολιτές δημοσιονομικού πλαισίου που δεν εγκρίθηκε καν ακόμα. Ευχαριστούμε κυρία Κιλέρα. Ευχαριστώ. Έχω κάποια σχόλια. Σίγουρα συμφωνώ με τους συναδέλφους σε πολλά σημεία. Πάλι προσπαθεί να μας πιέσει και να μας βάλει το μαχαίρι στο λαιμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε να κάνουμε κάποια στοιχεία του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη τι τελική μορφή θα έχει αυτό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αυτό θα καθορίσει και το πρόγραμμα των εργασιών γιατί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να καθορίσει τη θέση του, αλλά και γι' αυτό περιμένει το ΠΔΕΛΤΑΠΗ. Αλλά ε, προς τι αυτή η σπουδή λοιπόν, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Μετά τη μεταρρύθμιση του 92, αυτή είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Οπότε, προς τι αυτή η βιασύνη. Θέλω να μου διευκρινίσετε κάποια σημεία. Για παράδειγμα, το 2021 πώς θα χειριστούμε τις ενισχύσεις στα PDR. Όσοι έχουν ε, πόρους διαθέσιμους θα τους χρησιμοποιήσουν και τι θα γίνει με όσους δεν έχουν άλλους πόρους. Χρειαζόμαστε νέους πόρους. Στην πατρίδα μου την Ισπανία τα προγράμματα αυτά είναι περιφερειακά. Δεν τα διαχειρίζεται η κεντρική διοίκηση. Και στην Ιταλία και στη Γερμανία το ίδιο συμβαίνει. Αυτά τα προγράμματα είναι στα χέρια της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, όχι της κεντρικής κυβέρνησης. Οπότε χρειάζονται νέα κονδύλια σε περίπτωση που εξαντληθούν τα προηγούμενα. Είναι πολλά θέματα που θα πρέπει να ρυθμίσουμε. Και γι' αυτό χρειάζομαστε περισσότερο χρόνο. Συμφωνώ λοιπόν με τους συναδέλφους. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Ευχαριστώ, κυρία Λίεβα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι οι συνάδελφοι έκαναν σημαντικές ερωτήσεις. Εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη. Υπάρχουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις εδώ που κατά τη γνώμη μου δεν είναι ε, πλήρης. Ε, οι κρατικές ενισχύσεις ε, υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη οι ε, ε, ε, ορισμένες είναι και προσωρινές, ιδιαίτερα για την κτηνοτροφία. Εκεί θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και πώς θα διατηρηθούν, γιατί υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξαρτώνται πάρα πολύ από τις βοήθειες αυτές και το εισόδημα ορισμένων γεωργών κινδυνεύει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Κατάινεν. Στην Ευρώπη έχουμε 8 εκατομμύρια γεωργούς ε, που χρειάζονται σαφείς κανόνες και σαφή νομοθεσία από εμά για να κανονίζουν την πορεία τους, το μέλλον τους και τις επενδύσεις τους. Χρειάζεται σταθερότητα ο κλάδος. Και στη νέα ΚΑΠ τα πράγματα είναι πάρα πολύ θολά και συγκεχημένα. Ε, υπάρχει το πολιετές νομ, ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο, δημοσιονομικό, ε, που επίκειται και οι αγρότες χρειάζονται ένα αρκετά μεγάλο μεταβατικό διάστημα ε, για να μην δυσκολευτούν και να μην δυσκολευτούν και τα κράτη-μέλη από τις περικοπές. Χρειάζεται χρόνος για να γίνεται η νομοθεσία δεν ξέρω κατά πόσο αρκεί ένα έτος ε, ως μεταβατική περίοδος. Ευχαριστώ. Επόμενος συνάδελφος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, ο κύριος Χίτσβέγγι. Καλωσορίζω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τα δύο θέματα. Νομίζω ότι η σταθερότητα και η συνέχεια οικονομική είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως ακούσαμε προηγουμένως. Ε, μήπως θα είχε νόημα να τα δούμε χωριστά. Τώρα ε, καλά ε, τα έχετε παρουσιάσει από κοινού, αλλά για την ευελιξία για το 2020 πρέπει να λάβουμε γρήγορα απόφαση, ενώ για το άλλο, για το μεταβατικό διάστημα έχουμε χρόνο. Για το μεταβατικό κανονισμό, το δεύτερο, χαίρομαι που ε, επιτρέπουν ε, οι διατάξεις να έχει συνεχιστεί το σχήμα πληρωμών του ενιαίου χώρου. Δηλαδή ε, να υπάρχει μεταφορά πόρων από τον ένα πυλώνα στον άλλο. Να έχουν κάποια ευελιξία τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τα πολιετή μέσα. Παρόλα αυτά δεν είμαι πεπισμένο ότι το ένα έτος που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρκετό διάστημα για να γίνουν όλα αυτά. Το ανέφεραν πολύ προλαλήσαντες. Τα κράτη-μέλη χρειάζονται χρόνο για να αναπτύξουν τα στρατηγικά του σχέδια. Μετά χρειάζεται χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τα αξιολογήσει, να τα επιστρέψει στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ χρονοβόρο. Και για μένα δεν φτάνει ο ένας χρόνος. Είναι πολύ λίγο, μικρό διάστημα. Από την άλλη, ε, εγώ θα ήθελα να συνεχιστεί η ε, δυνατότητα χορήγησης κρατικής ενίσχυσης σε μεταβατική βάση. Αυτά δεν είναι κονδύλια που βαρύνουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά τον κρατικό της κάθε χώρας. Και είναι καλό για τον κλάδο, υπάρχουν και ευαίσθητοι τομείς και ερωτώ γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να σταματήσει. Ε, έγινε το 2014 θα ήθελα να συνεχιστεί και για το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ κυρία Βίνα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου πρόεδρε. Έχουν υποθεί όλα ουσιαστικά ε, δύο λεπτομέρειες για να δούμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η ομπρέλα για την οποία συζητάμε και να μην περάσουν όλα άρον-άρον. Ας πούμε συγκεκριμένα τι γίνεται με τις νέες υποχρεώσεις για την ε, ε, γεωργία για ε, το περιβάλλον, για το δεύτερο πυλώνα, για τα δάση κτλ. Προβλέπεται μία τριετία. Μα η οικολογική γεωργία χρειάζεται χρόνο για προσαρμογή και το Ταμείο Προσαρμογής προβλέπει πενταετία δεν θα ενισχύσει την αποδοχή του κοινού. Το δεύτερο, στην αιτιολογική σκέψη 28 λέει για να πάμε προς μια πιο δίκαιη κατανομή κουλουπού κουλουπού, δεν θα σας τα διαβάσω όλα, ε, ε στο επίπεδο του 2019 για την καταποκοπή καταβολή χρειάζεται ε, να ξεκαθαρίσουμε ε, τι γίνεται με τις περιφέρειες. Μα γιατί τα κράτη-μέλη μπορούν να κρατήσουν το 2021 τις δαπάνες σε επίπεδο του 2019 αντί να συνεχίζουν τη διαδικασία σύγκλησης των περιφερειών τους. Κύριε Καβαγιές, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, χαιρετίζω την πρόταση κανονισμού που είναι εντελώ κατεπήγουσα, αλλά μόλι τώρα μας έρχεται και δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να μπορέσουμε να τα μελετήσουμε κατά λεπτός. Ε, ερμηνεύοντας τις αυτές, ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να προσφέρουμε και κάποια... να καθησυχάσουμε τους ε, γεωργού και εκτινοτρόφους μα, αλλά να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρξει και σταθερότητα μετά τη μετάβαση. Για τις τιμές μάλιστα, τι προσωρινές του του δημοσιονομικού πλαισίου, ακούστηκε ήδη το σχόλιο, δεν είμαστε βέβαιοι. Και επίσης δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι για την πρόταση αυτή της εξωτερικής σύγκληση που χρειάζονται μεγαλύτερα αποθέματα και που δεν χρειάζεται εδώ να τις αναπτύξω περαιτέρω γιατί δεν έχουμε χρόνο, αλλά οι τιμές για το πρόγραμμα ΠΟΖΕΙ, ας πούμε, ε, δεν ακολουθούνται και πολύ σωστά. Και το έχουμε πει επανειλημμένως και στον πρόεδρο Γιούνκερ και στον επιτροπό Χόγκαν ότι θα πρέπει να σκεφτείτε τις ιδιαίτερα μειονεκτούσες περιοχές. Αυτές που έχουν ε, δομικές ε, μειονεξίες, αξιπέραστες ανυπέρβλητες μάλλον. Ε, πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν το θέμα αυτών των αποθεμάτων, ε, διότι εφόσον περικοπούν θα έχουν δραματικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές. Αυτές οι ενθερμό τρεις πρώτες αντιδράσεις και βεβαίως θα ήθελα απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσα είπα. Ευχαριστούμε κυρία Τολγαϊ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κείμενο αυτό που ε, λίγο το τελευταία στιγμή μας το στείλατε ε, με την επιφύλαξη μιας πιο ενδελεχούς μελέτης του κειμένου υπάρχουν ήδη κάποια σημεία τα οποία ήδη μπορούμε να τα πιάσουμε και να τα σχολιάσουμε. Πολύ αισιόδοξο να έχουμε μόνο ένα χρόνο μετάβαση ε, του σημερινού συστήματος Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, εφόσον συμφωνήσουν, θα πρέπει να προβλέψουν αρκετό χρόνο στα κρατη να συντάξουν τα στρατηγικά του σχέδια και μετά να τα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο των σημερινών δηλαδή συζητήσεων, να πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε σε διαθεσμική συμφωνία στα τέλη του 2020 είναι μάλλον απίθανο. Τα κράτη-μέλη επίση πρέπει να έχουν αρκετό χρόνο για να μπορέσουν να προετοιμάσουν τα στρατηγικά του σχέδια και να μην υπάρξουν καθυστερήσει στην εφαρμογή των διαφορών παρεμβάσεων. Έχουμε μια αρκετά οδυνηρή εμπειρία από το πρόγραμμα ανάπτυξη τη υπαίθρου και την υλοποίησή του. Κρατά στο μέλλον λοιπόν να μην έχουμε τόσο μεγάλη χρονική απόκληση, ακριβώ επειδή δεν προβλέψαμε αρκετό χρόνο για να προετοιμάσουν οι άνθρωποι τα προγράμματά του. Θα πρέπει οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να μπορούν να ε, κανονίσουν τι κινήσει του με αρκετό ε, περιθώριο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιτρέψουμε μια πραγματικά σωστή υλοποίηση όλων των μέσων υποστήριξη που προσφέρει η ΚΑΠ. Και επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε και για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και ότι βασίστηκε στι ε, τιμέ που ήδη είχε προτείνει. 5% μείωση σε ονομαστικού όρου ε, για την ΚΑΠ. Ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν για τη μεταβατική περίοδο, γιατί να προβλέψουμε αυτέ τι επιδοτήσει από την πλευρά τη ΚΑΠ. Θα συνεχίσουμε να σπιζόμαστε τον προπολογισμό που θέλαμε για το ερχόμενο διάστημα του Πουδουπού και επίση ο Επίτροπο Χόγκαν έχει δεσμευτεί για το πρόγραμμα αποζήτηση και την ε, διαφύλαξη του προπολογισμού του. Να διαφυλαχθεί και στη μεταβατική περίοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, αν γίνεται να παραμείνετε στο χρόνο ομιλία σας, ο κύριος... Ε, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το είπε και ο κύριο Χόσλιν, δεν ξέρω αν μπορώ να το υποσχεθώ και εγώ, ότι θα προλάβουμε, δεν θα προλάβουμε σε ένα χρόνο και δεν θα προλάβω και στο χρόνο που μου δίνεται. Το φως δεν θα πέσει τώρα από ό,τι φαίνεται. Ε, πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε λίγο την ιδέα του κανονισμού νη συν ένα. Ένα συν Ε, θα χρειαστούμε δύο, ε, εν συν δύο, θα πρέπει να χρειαστούμε τουλάχιστον δύο χρόνια μετάβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί είχαμε πει δύο χρόνια, εσεί λέτε τώρα ένα για την μετάβαση. Ε, ξέρουμε από την πράξη ότι συνήθω υπάρχουν περισσότερε καθυστερήσει. Και μετά είπατε παλιά μετερρύθμιση νέο χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι επιτρέπεται μια παράταση της μεταρρύθμισης, πράγμα που μπορεί να έχει και κάποια μειονεκτήματα όμως, γιατί θα πρέπει να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και επίσης αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν η μεταρρύθμιση αυτή ήταν σωστή. Ε, παλιά μεταρρύθμιση με απλώς ε, παράταση και νέα ποσά, φρέσκο χρήμα. Και τρίτη παρατήρηση, στην Γεωργία έχουμε πολλά προγράμματα πενταετούς διάρκειας. Μπορούν απλώς να παραταθούν Δηλαδή μόλις εκπνεύσουν στα 5 χρόνια μπορεί να πάνε στα 6 και στα 7. Είναι τόσο απλό. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σαντέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι με κάλυψαν σε πολλά σημεία. Θα ήθελα πάντως να επιμείνω σε δύο συγκεκριμένα θέματα. Καταρχήν, στη διάρκεια της παράτασης του προγραμματισμού κατά τη γνώμη μου δεν αρκεί ένας χρόνος, δεν είναι και πολύ ρεαλιστικό, γιατί αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τον Ιανουάριο του 2021 τα στρατηγικά του σχέδια για να τεθούν σε ισχύ το 2022. Δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έχουν κολλήσει και θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστεί ΚΑΠ ε, επιτόπου, ο ένας χρόνος μόνο παράταση μου φαίνεται μη ρεαλιστικός. Δεύτερο, όπως επισήμαναν οι συνάδελφοι, τι γίνεται με τον προπολογισμό για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΣΕΙ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι δεσμεύσεις που αναλύθηκαν από τον πρόεδρο Γιούγκερ αλλά και από τον Επίτροπο Γεωργίας τον κύριο Χόγκαν θα πρέπει να τηρηθούν και θα πρέπει να ανακτήσουμε τα κονδύλια του ΠΟΣΕΙ, να επαναφέρουμε τον προπολογισμό του προγράμματο αυτού για τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ροπέ τώρα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε για το τι θα συμβεί το 2021. Αλλά αν δεν λάβει χώρα το Brexit, θα χρειαστούμε και άλλες μεταβατικές περιόδους. Γιατί ποιο είναι το βασικό πρόβλημα τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι το Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αν δεν θεσπιστεί το πι, εμείς μένουμε με τα χέρια δεμένα. Είδαμε μία παράταση κατά ένα χρόνο μέχρι το 2020, αλλά τι θα γίνει, θα ξεκινήσουμε το 2021, την περίοδο 2021-2027 και πώς θα τη χρηματοδοτήσουμε. Ακόμη και παρατείνουμε την προηγούμενη περίοδο, δεν έχουμε αρκετά κονδύλια με μία απλή παράταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μεταφορά, αλλά δεν έχουμε συμφωνήσει σε αυτό. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει στις προτάσεις περικοπές στα γεωργικά κονδύλια, με, τα οποία, με τις οποίες δεν συμφωνούμε. Και θα δεχτούμε την υβριδική πρόταση που μας κατέθεσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να συμφωνήσουμε δηλαδή ουσιαστικά έμεσα και στις περικοπές που προτείνει για το γεωργικό προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι άδικη στη συμπεριφορά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για το σύνολο του προγράμματος και έτσι το κατατεμαχίζει ελπίζοντας ότι θα συμφωνήσουμε με τα κλάσματα του προγράμματος. Όχι, το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και χρειάζεται πολύ χρόνος για να εγγύψουμε στο θέμα αυτό διεξοδικά. Θα είναι σημαντική πρόκληση για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπούντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι αγρότες μας χρειάζονται σταθερότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα και δημοσιονομική σταθερότητα. Θα πρέπει να ξέρουν τι κονδύλια να περιμένουν για το μέλλον. Αν θυμάμαι καλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάστηκε 8 μήνες για να αποφανθεί για τα εθνικά στρατηγικά σχέδια. Οπότε δεν είναι αρκετή η παράταση κατά ένα χρόνο. Θα πρέπει ε, η παράταση να είναι τουλάχιστον διετής. Βέβαια, αν ολοκληρωθεί νωρίτερα η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, τόσο το καλύτερο. Αλλά οι αγρότες σήμερα θα πρέπει να ξέρουν α, η ενίσχυση θα δικαιούνται. Και αν ξέρουν ότι η ενίσχυσή του σήμερα είναι χ, να ξέρουν ότι η ίδια ενίσχυση θα ισχύει και θα είναι κατοχυρωμένη και την επόμενη διετία. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Έχουμε πολλές περικοπές στον προϋπολογισμό. Οι συνάδελφοι που είναι κατά τον περικοπών στον προϋπολογισμό τι θα κάνουν, θα ασκήσουν πιέσεις στις κυβερνήσεις τους για να μην γίνουν περικοπές. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερες δράσεις με λιγότερα χρήματα. Και στη Γεωργία μπορούμε να έχουμε κάποια κρατικά κονδύλια για τη στήριξή της, αλλά φαίνεται ότι γίνονται περικοπές και στα κρατικά κονδύλια. Επιτρέψτε τουλάχιστον στα κράτη-μέλη να βοηθήσουν εκεί που χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σχρέιρ Πίρικ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σύντομα. Το είπε και ο κύριος Μπούντα τώρα μου. Φανταστείτε να είσαι αγρότης ή αγρότησα και να ακούς αυτή τη συζήτηση και θες να επενδύσεις στο μέλλον σου. Είσαι νέος αγρότης και σου λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνεις και πράγματα για το κλίμα. Μα τι θα κάνεις τι συζητάμε όλοι. Έχουμε ένα τεράστιο ε, χρέος και ευθύνη το συντομότερο να συμφωνήσουμε και να μην αναλωθούμε τους επόμενους μήνες ε, στην ε, σχολαστική ενασχόληση με αυτό το θέμα και να ψάχνουμε την κάθε γωνιά. Και στη χώρα μου. Με αυτό ασχολούνται με τα στρατηγικά σχέδια και τι θα κάνουμε θα πρέπει να δείξουμε μια πειθαρχία και να προχωρήσουμε ε, γρήγορα. Αυτή την έκκληση πραγματικά ήθελα να την κάνω. Ευχαριστώ, η κυρία Σμιτμπάου. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Και από τη σκοπιά των Αυστριακών αγροτών και αγροτησών πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να βιαστούμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτα είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από την άλλη ε, οι άνθρωποι, έτσι να το σκεφτούμε. Ε, σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν άνθρωποι με το πεπρωμένο τους και ακούσαμε ότι εξαφανίζονται διάφορα είδη, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εξαφανίζονται και αγρότες και θέλω να χάσουμε όσο γίνεται λιγότερους. Για την επιμήκυνση και παράταση των προγραμμάτων έχω μια ερώτηση και σας παρακαλώ πραγματικά να μου την απαντήσετε. Πολύ απλό ακούγεται αυτό. Παρατείνουμε μεταβατικές περίοδοι. Ποιες θα είναι όμως οι προϋποθέσεις για την παράταση. Πολύ απλό μου φαίνεται και δεν μπορώ να το φανταστώ τόσο απλό. Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις για την παράταση, ποια θα είναι τα κριτήρια ε, για να καταθέσει κανείς αίτηση παράτασης και θα εγκρίνονται κιόλα οι αιτήσει αυτές. Ευχαριστώ. Εξαντλήθηκε ο κατάλογος των ε, ερωτήσεων. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο και θα ξαναδώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγιναν μια σειρά ερωτήσεων και διαπιστώσατε κι εσείς ότι χρειάζεται πολύ συζήτηση. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και για όλες τις ερωτήσεις σας και τα σχόλια. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσες γίνεται περισσότερες. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας να σας εξηγήσει όλα τα θέματα, γιατί ορισμένα μπορεί να σας φαίνονται πολύ τεχνικά ε, και όπου θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε σε όποιο φόρουμ. Ε, ευχαριστώ. Ε, είμαι ευγνώμων σε όλους όσοι μιλήσατε υπέρ του διαχωρισμού των δύο προτάσεων. Από τη μια έχουμε τον κανονισμό για την ευελιξία που είναι πραγματικά κατεπήγον και θα πρέπει γρήγορα να εγκριθεί και κατανοούμε και χαιρόμαστε ότι χρειάζεται ε, βαθύτερη συζήτηση και περισσότερο χρόνο, άλλο ο κανονισμό για τη μεταβατική περίοδο και προσβλέπουμε στη συνεργασία το επόμενο διάστημα. Να δανειστώ το παράδειγμα από το 2013 και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρότεινε ένα μεταβατικό κανονισμό τον Απρίλιο, ο οποίο συμφωνήθηκε στο τριμερή διάλογο από του συνομοθέτε τον Οκτώβριο. Γίνονται λοιπόν αυτά τα πράγματα και πάνω κάτω ήταν οι ε, ίδιοι κανόνες και η ίδια περιπλοκότητα και κατάφεραν όμως οι συνομοθέτες να το χειριστούν ε, με μεγάλο επαγγελματισμό και ε, σε βάθος. Τώρα, για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, από την αρχή θέλω να πω ότι δεν προεξοφλούμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Δεν ήταν καθόλου η πρόθεση αυτής της πρότασης. Αλλά δεν μπορούσαμε να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για το PDP για τους λόγους που και εσείς αναφέρατε. Ότι είναι σχετικά αργά ήδη. Το καταλαβαίνουμε. Τι να κάναμε τώρα, να περιμένουμε άλλους τρεις-τέσσερις μήνες. Ε, ε, δεν θα μπορούσαμε να κενήσουμε τη διαδικασία ε, συνομοθέτησης και δεν ε, είχε συμφέρον κανείς ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιμένει να συμφωνηθεί το PDP για να φέρουμε την πρόταση. Αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε ένα ορόσημο που είναι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ταυτόχρονα όμως έχουμε υπόψη μας ότι αυτό ενδεχομένως δεν θα είναι και το τελικό κείμενο του PDP. Γι' αυτό είπα από την αρχή ήδη ότι όταν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα έχουν συμφωνήσει για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι λογικό και επόμενο και περιμένουμε όλα τα αριθμητικά στοιχεία και τα ποσά που έχουμε εδώ να αντικατασταθούν από τα νέα ποσά του ε, συμφωνηθέντος PDP. Ε, αυτό μπορεί να, να παρηγορεί λίγο τον κύριο Ντόρφμαν που λέει ότι έχουν μειωθεί πολύ τα κονδύλια ε, στο δεύτερο πυλώνα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Μα βλέπουμε ότι εκεί γίνονται συζητήσεις ε, που μας οδηγούν τελικά σε αύξηση ε, αυτού του πόρου. Ενδεχομένως λοιπόν οι περικοπές τις οποίες αναφερθήκατε να μην είναι τόσο οδυνηρές. Το δεύτερο και πάλι για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι το εξής εργαζόμαστε εμείς ε, με την εξή βάση. Ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα συμφωνήσουν για το PDP πριν υπάρξει η οριστική συμφωνία για το μεταβατικό μας κανονισμό. Αυτή ήταν η αρχική μας υπόθεση. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή στην τελική συμφωνία για το πολιετές, προτείνουμε ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το προσαρμόσει στη συνέχεια. Νομίζω ο κύριος Ντόρφμαν και ο κύριος Χόισλινγκ ρώτησαν τι γίνεται με τα προγράμματα στα κράτη-μέλη ε, που είναι αποκεντρωμένα. Ε, μα το έχουμε λάβει υπόψη αν δείτε την πρόταση. Υπό ποια έννοια. Τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νέο χρήμα με τους παλιούς κανόνες. Αυτή τη στιγμή έχουν εξαντλήσει τα παλιά κονδύλια. Αυτό εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη που έχουν ένα εθνικό σχέδιο. Για εκείνα τα κράτη-μέλη που έχουν περιφερειακά σχέδια, αυτό θα εφαρμοστεί σε επίπεδο περιφέρειας. Ας πούμε, Γερμανία και Ιταλία θα δούνε ποια από τα περιφερειακά τους προγράμματα έχουν ήδη εξαντληθεί εκ των παλαιών και από αυτές τις περιφέρειες ε, θα υπάρξει νέο χρήμα που θα δαπανηθεί με τους παλιούς κανόνες. Μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση, θα υπάρξει. Ε, Το επόμενο θέμα που θέσατε ορισμένοι από εσάς είναι οι μεταβατικές, οι προσωρινές κρατικές ενισχύσεις. Είναι γεγονός ότι στην πρότασή μας δεν προτείνουμε να παραταθεί αυτό. Μπορώ να σας εξηγήσω σύντομα για ποιο λόγο. Το λέει ο λόγος, γιατί υποτίθεται ότι ήταν προσωρινή η μεταβατική αυτή η βοήθεια. Το 2013 αποφάσισαν να παραταθεί μέχρι το 2020 αυτή η ρύθμιση και μόνο μέχρι το 2020. Συνεπώς, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση δεν προβλέπει συνέχιση αυτής της προσωρινής μεταβατικής ενίσχυσης μετά το 2020 και σεβόμαστε την ίδια μας την πρόταση που είπαμε ότι σταματάμε το 2020 και δεν έχουμε περαιτέρω παράταση. Έγινε και μια ερώτηση νομίζω από την κυρία Βίνερ για την εσωτερική σύγκληση και την ευελιξία που θα έχουν ε, τα κράτη-μέλη, θα τους εγκρίνουμε αν ακολουθήσουν αυτή την πρόταση. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο αυτό σε κάποια κράτη-μέλη και είναι ένα θέμα που συζητήθηκε και στην ίδια την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Λοιπόν, δίνουμε τις εξής δύο δυνατότητες στα κράτη-μέλη. Όσοι θέλουν να συνεχίσουν στην εσωτερική σύγκληση ε, να επιτραπεί να το κάνουν και μετά το 2020-2021. Και όσοι λέγουν όχι, θέλουμε να σταματήσουμε στο επίπεδο του 2019 που είναι το τελευταίο έτος με τους παρόντες κανόνες, μπορούν να σταματήσουν το ρολόι ας πούμε και να δούμε τι θα αποφασίσουν οι συνομοθέτες για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Επίσης, πολλοί ρωτήσατε για το πρόγραμμα ΠΟΣΕΙ και άλλα προγράμματα και τη χρηματοδότησή τους, εδώ δεν μπορούμε παρά να επαναλάβουμε ότι αυτό που κάνουμε στην πρότασή μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε τα ποσά από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το PDP και τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, γιατί μόνο αυτή την αναφορά έχουμε. Εάν αλλάξουν τα πράγματα όσο προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, βεβαίω θα ε, βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα το 2021. Ο κύριος Γιάρ, νομίζω, ανέφερε κάτι για το νησιν 2 σε σχέση με το νησιν 3 οι τρέχοντες κανόνες για ε, τα παλιά κονδύλια προβλέπουν τον ίσιν 3. Αυτό δεν αλλάζει. Για τα κράτη Κίνα όμως που θα παρατείνουν τα προγράμματά τους ανάπτυξης υπαίθρου ε, το 2021 θα ισχύσει και πάλι ο κανόνας του νησιν 3. Το νησιν 2 θα είναι νέος κανόνας μόνο για τη μεταρρύθμιση και όχι για το μεταβατικό έτος. Εκεί ποντάρουμε στην συνέχεια στα πλαίσια και των άλλων προτάσεών μας. Ένα προτελευταίο σημείο. Τι γίνεται με την ε, ανάληψη υποχρεώσεων για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος και τη χρονική διάρκεια. Εκεί έχουμε ένα δίλημα. Αν δούμε πώς δεσμεύεται ο κάθε αγρότης, προφανώς ε, όταν είναι πιο μακράς πνοής, ε, είναι καλύτερο από ότι είναι βραχυχρόνιο. Αν το δούμε στρατηγικά όμως, τι θέλουμε να πούμε. Ότι να υπάρχουν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα ε, ελεύθερα για τα κράτη-μέλη ε, όταν αρχίσουν να εφαρμόζουν τα στρατηγικά σχέδια. Γιατί στόχος είναι να έχουν υψηλότερους στόχους, πιο στοχευμένη ενίσχυση ακριβώς για το περιβάλλον και το κλίμα και αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε μαζί με τους αγρότες σε ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Και όσο πιο μακροπρόθεσμα δεσμεύεσαι για 3, 5 ή 7 χρόνια, τόσο ακριβώς δεσμεύεσαι, δεν είναι στα χέρια σου και δεν έχεις τα χρήματα για να τα δαπανίσεις στα σχέδια τα στρατηγικά. Γι' αυτό είπαμε για το 2021. Στην ανάληψη υποχρεώσεων ε, προβλέπουμε από ένα έως τρία έτη για να μεγιστοποιηθεί το κέρδος ε, στα στρατηγικά σχέδια. Να έχουν τη δυνατότητα όσο μπορούν πιο ελεύθερα να δαπανούν τα κόντυλια αυτά. Και το τελευταίο θέμα, αυτό το, το ταμπού που δεν συζητάει κανείς, ε, ε, που είναι η διάρκεια το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2013, νομίζω τον Απρίλιο, αρχίσαμε τον τριμερή διάλογο και τον Ιούνιο είχαμε την τελευταία ε, πολιτική απόφαση. Όλα αυτά μπορεί να γίνουν σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ε, έτσι κάναμε και την πρότασή μας, ε, στηριζόμενοι στην εμπειρία του 2013. Και αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούν οι συνομοθέτες να καθίσουν, να διαπραγματευτούν του επόμενου μήνες, να αρχίσουν τριμερείς διάλογοι την Άνοιξη και ελπίζουμε να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τη μεταρρυθμίση αυτή καθ' αυτή περί το θέρο. Και οπότε έχει νόημα και ο περιορισμός σε ένα χρόνο, το 2021, αν υπάρξει καθυστέρηση, καταλαβαίνω ότι μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου. Αλλά σήμερα θέλω να σας απευθύνω την έκκληση. Ας δούμε πρώτα την ουσία της πρότασης και το χρονικό να το δούμε αργότερα. Όταν θα έχουμε περισσότερη σαφήνεια για το πού βρισκόμαστε, πώς πάει η διαδικασία μεταρρύθμισης, ε, γύρω στο, στην άνοιξη το καλοκαίρι του 2020. Σας ευχαριστώ πολύ. Ja, vielen herzlichen Dank. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τις διεκθρωτικές απαντήσεις. Προφανώς το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας ξανά και ξανά και μπορείτε να μεταφέρετε στον Επίτροπο ότι δείξαμε την διάθεση εμπιστοσύνη μας να επιταχύνουμε την έγκριση του κανονισμού ε, ευελιξίας. Αλλά για τη δεύτερη πρόταση η Επιτροπή ετοιμαστεί για περισσότερες συζητήσεις. Πείτε τα αναλόγως και στον Επίτροπο. Συνάδελφοι, φτάσαμε στο τέλος της ημερήσιας διάταξης και το τέλος του σημείου 11. Οπότε πάω απευθεία στο 12. Έγκριση των συστάσεων των συντονιστών της Επιτροπής Άγκρη, αυτές που λάβαμε νωρίτερα το πρωί, σας έχουν αποσταλεί. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνονται. Πάμε λοιπόν στο σημείο 13, διάφορα. Υπάρχει κάτι στα διάφορα από πλευρά σας. Ο συνάδελφος Γιούργελ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την απάντηση στην ερώτησή μου που διέφυγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέφυγε μάλλον απαντήσει, να μου την απαντήσει γραπτός, παρακαλώ. Εννοείται την ερώτησή σας προηγουμένως. Στην προηγούμενη συζήτηση, στο προηγούμενο, προ-προηγούμενο σημείο της Μέσας Διαταξής. Ναι, εντάξει. Υπό τα διάφορα κάτι άλλο, παρακαλώ, κυρία Αγγιλέρα. Ζητώ συγγνώμη κάτι για τις στάσεις των συντονιστών. Ε, μου λέει ο συντονιστής μας ότι στην αποστολή, στην Εστρεμαδούρα, στην Ισπανία, ε, προβλέπεται για το επόμενο εξάμεινο, το Μάιο. Τι συνιστούν όμως οι συντονιστές γι' αυτό. Δεν το βλέπω πουθενά. Μου λέει ο κύριος Δεκάστρο ότι συζητήθηκε, αλλά δεν το βλέπω πουθενά γραμμένο στις συστάσεις των συντονιστών. Για να το διευκρινίσω, ερωτώ. Συνάδελφε Αγγιλέρα, τα έχουμε ξανασυζητήσει, απλώς σήμερα δεν λάβαμε απόφαση. Αποφασίσαμε ότι θα γίνει ταξίδι στην Ισπανία, αλλά όχι τι λεπτομέρειε. Ούτε πού ακριβώς, ούτε περί τίνο θα πρόκειται. Συνάδελφε Ντόρφμαν, έχετε κάτι να πείτε κι εσείς. Αυτή είναι η κατάσταση όσο έχει τώρα. Γι' αυτό λοιπόν σύσταση των συντονιστών είναι να ληφθεί απόφαση, διότι ακόμα δεν έχουμε καταλήξει οριστική απόφαση. Ε, ε, Δεκάστρο, μα νομίζω η απόφαση ελήφθη, Πρόεδρε. Είπαμε Μάιο, Ισπανία. Και είπαμε ότι απλώς θα είναι αποστολή σε κάποια περιοχή της Ισπανίας. Νομίζω ότι η απόφαση έχει ληφθεί. Τι να περιμένουμε άλλο. Ακριβώς. Αυτό αποφασίσαμε. Όχι το περιεχόμενο όμως της απόφασης όχι πού ακριβώς θα πάμε, αν θα βρούμε κάποια συμβαστική λύση, ποια από τις δύο περιοχές, ε, πού θα είναι ο προορισμός μας, αυτό δεν έχουμε αποφασίσει. Άλλες παρατηρήσεις στα διάφορα, άλλος κατάλαβε διαφορετικά την απόφαση. Κύριε Αγγιλέρα, η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς ως σοσιαλιστική ομάδα είναι να πάμε στην περιφέρεια της Εξτρεμαδούρα. Είναι μία πρόταση μοναδική Ποιε είναι οι, δεύτερες, οι δύο περιφέρειες, υπάρχει άλλη πρόταση από άλλη ε, πολιτική ομάδα. Η πρόταση δεν ήταν να πάμε σε δύο περιφέρειες. Εμείς κάνουμε μία πρόταση ως πολιτική ομάδα και σας το λέω για να το διευκρινίσουμε. Πρέπει να ληφθεί απόφαση ξεκάθαρη. Ό,τι και να αποφασιστεί, να ξέρουμε τι θα κάνουμε και πού θα πάμε. Η πρόταση των σοσιαλιστών και δημοκρατών είναι Ισπανία-Εξτρεμαδούρα. Genau. ne? Ακριβώς. Επαναλαμβάνω. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, κύριε Ντόρφμαν. Πρόεδρε, έχεις δίκιο. Αποφασίσαμε στη συνεδρία των συντονιστών να πάμε στην Ισπανία και την Ουγγαρία. Μέχρι εκεί. Αυτή η απόφαση έχει ληφθεί. Από εκεί και πέρα θα πάρουμε προτάσεις για τα προγράμματα που στις χώρες αυτές υπάρχει κάτι ενδιαφέρον να πάμε να δούμε. Αυτό θα το αποφασίσουμε. Αυτή τη στιγμή δούμε και τα αντίστοιχα προγράμματα. Άλλε παρατηρήσει υπό τα διάφορα για αυτό το θέμα, για κάτι άλλο, όχι. Πάμε στο 14, η επόμενη συνεδρίαση στις 18 Νοεμβρίου και μετά 4 και 5 Δεκεμβρίου με τις σχετικές ακροάσεις. Σας εύχομαι καλή, καλό βράδυ. Θα τα πούμε το αργότερο μέχρι στην επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστούμε.